comenzamos nuestra audición sobre la libertad de expresión y la democracia en Hong Kong. Los anuncios que como presidente. Λοιπόν, τις ανακοινώσεις της Προέδρου θα τις κάνω αργότερα γιατί έχουμε συγκεκριμένο ωράριο για τη σύνδεση με βίντεο με τους ομιλητές που θα πρέπει να ε, συζητήσουν μαζί μας με βάση τα πρόσφατα γεγονότα όλοι γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν σοβαρά πράγματα στο Χονγκ και θα θέλαμε να μάθουμε απευθείας τη γνώμη των ατόμων που ζουν εκεί. Τα γεγονότα αυτά συμβαίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και γι' αυτό δύο από τους εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές που προσκαλέσαμε προτίμησαν να μείνουν στο Χονγκ και να μας μιλήσουν από εκεί. Το πρώτο λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να έχουμε μια ε, κατά το δυνατόν ευρύτερη θεώρηση του τι συμβαίνει, ούτως ώστε μετά, εάν χρειάζεται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημοκρατίας και την εγκαθίδρυση της ελευθερίας έκφρασης στο Χονγκ είναι θέμα που σχετίζεται άμεσα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και αυτό είναι θέμα ενδιαφέροντος και αρμοδιότητας της Επιτροπής μας από πλευράς θεσμικής και ε, γι' αυτό ε, θέλουμε να έχουμε διάλογο και με τις ε, αρχές της Κίνας και του Χονγκ και γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει να μας μιλήσουν άτομα που έχουν συμμετάσχει στα γεγονότα Κάτι που συνέβη χθες καινούριο που θέλω να μας το σχολιάσουν. Διάβασα ότι τρεις καθηγητές που ηγούντο των ε, διαδηλώσεων ζήτησαν από τους ε, φοιτητές να σταματήσουν οι διαδηλώσεις και ότι οι τρεις αυτοί θα παραδοθούν στις αρχές για να αποφευθούν ε, περαιτέρω επεισόδια βίας όπως αυτά που συνέβησαν πρόσφατα. Ευχαριστώ επίσης την αντιπροσωπεία μας στο Χονγκ που μας διευκόλυνε για την διεξαγωγή αυτής της ακρόασης και τη γραμματεία της Επιτροπής μας που εργάστηκε ούτω ώστε σήμερα να έχουμε αυτή τη σύνδεση και την παρουσία της εμπειρογνώμονος της αρμόδιας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Χονγκ Κόνγκ που είναι εδώ και θα συντονίσει τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σύνδεση βίντεο, ούτω ώστε οι συνομιλητές μας να μπορέσουν να μιλήσουν αμέσως. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Λάου Ιουκάη, που είναι επικεφαλής ε, της ε, μη κυβερνητικής οργάνωσης ε, ανθρώπινα δικαιώματα στο Χονγκ Κόνγκ παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Χονγκ που συνεργάζεται και με τα Ηνωμένα Έθνη θα του ζητήσουμε να μας ενημερώσει για την άποψή του για τα γεγονότα των τελευταίων μηνών και να μας μιλήσει επίσης για το ενδεχόμενο μεταρρυθμίσεων θεσμικών και εκλογικών που θα βοηθούσαν κατά τη γνώμη του. Ελπίζω να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ κύριε ε, Λάου Ιουκάι, ε, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας ε, καλέσατε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Χονγκ Κόνγκ όπως επίσης και για το πόσο ανησυχείτε για τις δημοκρατικές εξελίξεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Human Rights Monitor είναι ε, μια μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο για την προστασία ε, των ε, οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Hong Kong. εδώ και 20 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε εκστρατεία υπέρ της δημοκρατίας διατηρούμε την ε, ε, δυνατότητά μας βάσει του άρθρου 9 ε, του Διεθνούς Συμφώνου για τα πολιτικά μας δικαιώματα και μιλάω ειδικότερα για το σημείο 34 και βάσει των αρχών του Johannesburg να προσπαθούμε να ε, συνεχίσουμε αυτό μας τον αγώνα. Η αστυνομία του Hong Kong ε, μας υποσχέθηκε να μας βοηθήσει και εμάς και τους δημοσιογράφους τον Ιούλιο του 2011. μέχρι πριν από 7 μέρες η αστυνομία ε, προσπάθησε ε, να παρεμποδίσει ε, και τους παρατηρητές αλλά και τους δημοσιογράφους και προσπάθησε επίσης να παρεμποδίσει ε, όλες τις προσπάθειές μας ε, για ε, διαδηλώσεις. χρειαζόμαστε καλύτερη λογοδοσία της αστυνομίας. Το ακόμα ε, το κίνημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει ε, στο Χονγκ Κόνγκ ε, αφορά την δυνατότητα ύπαρξης καθολικών εκλογών υπό ανεξάρτητη παρακολούθηση ανεξάρτητων παρατηρητών. Οι αρχές του Χονγκ Κόνγκ δεν προ, δεν ε, προκύπτουν από, ε, από καθολική ψηφοφορία. Ε, οπότε αυτή τη στιγμή η εκτελεστική εξουσία δεν ψηφίζεται απευθείας από το λαό του Χονγκ Κόνγκ και δεν υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση. υπάρχουν πολλά προβλήματα για διάφορους τομείς της κοινότητας η Επιτροπή Μελέτης ε, του Εθνικού Κογκρέσου ε, της Κίνας ε, το καλοκαίρι αποφάσισε ότι η εκλογή του κυβερνήτη του Χονγκ Κόνγκ το 2017 πρέπει να είναι αποτέλεσμα ψηφοφορίας ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Αυτό όμως υπόκειται στον περιορισμό ότι οι υποψήφοι πρέπει να ε, διορίζονται από την Επιτροπή ε, του Εθνικού Κογκρέσου της ε, Κίνας. Η Επιτροπή θα επιλέξει δύο με τρεις υποψηφίους και η πλειοψηφία τουλάχιστον, και με πλειοψηφία τουλάχιστον του ημίσεως της ε, Επιτροπής ε, της Αρμόδιας του Εθνικού Κογκρέσου της Κίνας. Οι άνθρωποι ε, λοιπόν οι οποίοι δεν εγκρίνονται από το Πεκίνο, αν δηλαδή το Πεκίνο δεν εγκρίνει κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν μπορούν να είναι υποψήφοι για τη θέση του κυβερνήτη. Και το Πεκίνο είναι αυτό που διορίζει τους συγκεκριμένους υποψηφίους. Αυτό αυτή λοιπόν, ε, οι, αυτές οι ψευδοεκλογές θα δώσουν την ε, επιλογή ε, μεταξύ κακών και χειρότερων υποψηφίων. Δεν είναι μια πραγματική επιλογή, δεν είναι μια πραγματική επιλογή για τον κόσμο. δεν είναι μια κυβέρνηση που προκύπτει από την πραγματική βούληση του λαού. είναι λοιπόν μια ψευδής εκλογή η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ε, ζητά το ζήτησε μια πραγματική εκλογική διαδικασία στις 26 Σεπτεμβρίου ε, και ε, έγιναν διαδηλώσεις μπροστά από ε, τις ε, εγκαταστάσεις της κυβέρνησης. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε καμία δυνατότητα πρόσβασης. Ήρθε, βγήκαν, βγήκαν στους δρόμους οι πολίτες από όλες τις γωνιές του Χονγκ Κονγκ. Δυστυχώς όμως υπήρξε καταστολή από τους αστυνομικούς. Κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι φοιτητές μάλιστα συνελήφθησαν στην πλατεία Δημοκρατία. Στις 28 Σεπτεμβρίου οι φοιτητές και πολλοί διαδηλωτές ε, ε, απομακρύνθηκαν από την περιοχή Κάποιοι προσπάθησαν μάλιστα να προστατέψουν τους φοιτητές και προσπάθησαν ε, ε, να χρησιμοποιήσουν διάφορες μάσκες ε, για να αντιμετωπίσουν ε, τα διάφορα αέρια που χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί οι φοιτητές. Μάλιστα ζητήθηκε από τους φοιτητές να σταματήσουν να να στεβαστούν την, ε, τις, ε, τις γραμμές, τις ε, λωρίδες της αστυνομίας. Η, η αστυνομία άρχισε να χρησιμοποιεί δακρυγόνα αέρια κατά των διαδηλωτών και μάλιστα ο διοικητής της αστυνομίας είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν τα δακρυγόνα ε, για να μπορέσουν να αποθήσουν τον κόσμο ε, όταν ε, ε, πλησίαζε την προστατευόμενη από την αστυνομία περιοχή. Όταν προσπάθησαν λοιπόν να αποθήσουν τον κόσμο πέρα από τις ε, λωρίδες αποκλεισμού της αστυνομίας. Δεν χρειαζόταν όμως να χρησιμοποιηθούν ε, δακρυγόνα, ούτε χρειαζόταν τόση βίαιη συμπεριφορά ε, κατά των διαδηλωτών. Μετά από χρήση πάρα πολλών δακρυγόνων, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά δακρυγόνα χωρίς να υπήρχε λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, προσπάθησαν ε, να χρησιμοποιήσουν ε, ε, διάφορα σπρέι δακρυγόνα ανεξαιρέτως κατά των διαδηλωτών και σε μερικές περιπτώσεις τέτοιου είδους ε, βία ε, χρησιμοποιήθηκε ακόμη και εναντίον ε, ιατρών που ήταν εκεί επιτόπου προσπαθώντας να παρέχουν ιατρική φροντίδα όταν χρειαζόταν και κατά δημοσιογράφων και άλλων παρατηρητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κάποιοι άλλοι ε, παρατηρητές ε, ε, σπρώχτηκαν, τοποθετήθηκαν στους τοίχους ασκήθηκε σωματική βία από τους αστυνομικούς. Ακόμη και περαστικοί ε, πολλές φορές ήταν ε, αντικείμενο επίθεσης χωρίς κανένα λόγο. Η αστυνομία ε, φαίνεται να έχει τον έλεγχο. Στις 15 Οκτωβρίου 7 αστυνομικοί συνέλαβαν υπόπτους, έναν ύποπτο, τον οποίο τον έριξαν στο πάτωμα, του έβαλαν χειροπέδες, τον γρομφοκόπησαν κατά συρροή και και κάποιοι μάλιστα το μαγνητοσκόπησαν. Ε, υπήρχαν ε, διαδηλωτές, ε, υπήρχαν άνθρωποι περαστικοί που τους χτύπησαν στην πλάτη χωρίς ε, να προβούν σε καμία προκλητική συμπεριφορά και μάλιστα αυτό ήταν κατόπιν εντολής αστυνομικού. Ε, τον, το να χρονθοκοπεί κανείς περαστικούς και διαδηλωτές ε, είναι πλέον κοινή πρακτική στο πλαίσιο των διαδηλώσεων αυτών στο Χονγκ Κονγκ. Ε, τι νόημα έχει... Χρησιμοποιεί κανείς κλόμπ στην πλάτη των ανθρώπων. είναι απλώς μια εκδήλωση οργής. Θέλω λοιπόν να κάνω την αξή ερώτηση. Σε ποια χώρα της Ευρώπης θα μπορούσε κανείς ε, να δεχθεί ε, να χρησιμοποιούνται κλόμπ από την αστυνομία ή τέτοιου είδους βία σαν αυτή που περιέγραψα ε, λόγω πίεσης, λόγω πολλών ορών εργασίας ή λόγω θυμού. Έτσι όμως έχουν τα πράγματα και οι παρατηρητές ε, μάλιστα ε, απομακρύνονται Είδαμε και άλλα είδη ε, βίας στις αρχές του Οκτώβρη μαφιόζοι από τις ε, τριάδες ε, επιτέθηκαν σε διαδηλωτές και πήρε πάρα πολύ χρόνο ε, η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων επιτόπου. Ε, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι δεν είχε κανένα νόημα η αστυνομική παρουσία. Η υπεύθυνοι αυτή της επίθεσης ε, συνελήφθησαν, οι ε, ε, ήδη διατηλωτές τους παρέδωσαν στην αστυνομία. Πολλέ φορέ όμω τους πήγαιναν στο μετρό και τους επέτρεπαν να φύγουν. Και Όταν κάποιος ας πούμε ήθελε να καταθέσει ε, εναντίον ε, αυτών των ε, ανθρώπων που έκαναν σε αυτές τις επιθέσεις, η αστυνομία δεν ενδιαφέρεται καθόλου. αν κάποιος ας πούμε έχει, έχει συλληφθεί και κρατείται χωρίς στοιχεία, μετά πρέπει να απελευθερωθεί. Αν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Τώρα είναι δύσκολη η κατάσταση υπάρχει καταστολή και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνουν συστάσεις για να ε, κάνουν έκκληση ε, προς τις ε, ε, αρχές ε, του ε, Hong Kong και της Κίνας να λύσουν το ζήτημα πολιτικά και όχι μέσω της βίας. Να μην χρησιμοποιείται βία, να μην χρησιμοποιούνται τα GLOBE ως βασικό τρόπο συμμόρφωσης των διαδηλωτών. Να μην χρησιμοποιείται λοιπόν η βία κατά των διαδηλωτών, κατά των παρατηρητών και κατά των διαδηλωτών και κατά των δημοσιογράφων. Και όσοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίζουμε να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ του Πεκίνου ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικό αυτό το πρόβλημα ε, που υπάρχει στο Χονγκ Κόνγκ. Παρά το γεγονός ότι μας έχουν υποσχεθεί μία χώρα και δύο συστήματα, ε, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες στο Χονγκ Κόνγκ είναι συνεχώς υπό απειλή και κυρίως η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθε. Υπήρξαν πάρα πολλέ ε, συλλήψει, άνευ προηγουμένου είναι ο αριθμός κατά τα πρόσφατα ε, χρόνια. Και για την ελευθερία της έκφρασης, το βασικό είναι η λογοκρισία στο ίντερνετ. Υπάρχει παρέμβαση από τις, ε, κοινωνικές αρχές, τις κινέζικες αρχές και υπάρχει επίσης και νομοθεσία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς το συμφέρον των κινέζικων αρχών. Σύμφωνα με ερευνητές, η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς οι ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις είναι αυτές ε, που η ε, ραδιοτηλεόραση είναι αυτή η οποία ε, υποφέρει περισσότερο ως προς την ανεξαρτησία της. Υπάρχουν χειρότεροι τρόποι κανείς να ασκήσει πίεση όσον, για παράδειγμα μέσω της ε, ανανέωσης της άδεια λειτουργίας αυτών των μέσων ενημέρωσης. Η κυβέρνηση προσπάθησε μάλιστα να παρεμποδίσει και την έναρξη λειτουργίας ενός νέου φορέα και πάρα πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ε, για να διαδηλώσουν κατά της ε, απαγόρευσης λειτουργίας ε, μιας τοπικής ραδιοτηλεόρασης. Επίσης είδαμε πολλά προβλήματα με την δημόσια ραδιοτηλεόραση γιατί η κυβερνητική παρέμβαση είναι μεγάλη. Είναι αδύνατον η δημόσια ραδιοτηλεόραση να διεκπαιρεώσει το ρόλο της με ανεξάρτητο τρόπο. Σας ενημερώνω λοιπόν για όλα αυτά τα προβλήματα θα ήθελα να ληφθούν υπόψη ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πραγματική δημοκρατία στο Χονγκ Κόνγκ πώς ε, έχει προβλεφθεί στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ε, πολιτικά δικαιώματα και βασικές ελευθερίες όπως τις ελευθερίες και του συνεταιρίζεστε να την χάνουν πραγματικής προστασίας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εδώ επίσης το καθηγητή Wong Wai Kok Benson από το Τμήμα Διεθνών Σπουδών του Βαπτιστικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κόνγκ συμμετέχει ε, σε ένα πρόγραμμα που ε, ονομάζεται Μετάβαση στο Χονγκ Κόνγκ, δηλαδή ε, η διαδικασία μετάβασης του Χονγκ Κόνγκ και έχει συνεργαστεί με διάφορες οργανώσεις νεολαίας στο Χονγκ Κόνγκ. Οπότε νομίζουμε ότι έχει πολλή έννοια να μας μιλήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε η δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας το τι ακριβώς συμβαίνει στο Χοκόγκ. Ο προηγούμενος ομιλητής ανέφερε ορισμένα στοιχεία των όσων συμβαίνουν στο Χονγκ και αναφέρθηκε και, και στις επιθέσεις των αστυνομικών δυνάμεων, τις δειλές ε, ε επεμβάσεις, καθώς ε, και το γεγονός ότι καλείται η κυβέρνηση να δώσει μια απάντηση στα δημοκρατικά αιτήματα του λαού του Χονγκ Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια παρατήρηση με βάση αυτές τις ιδέες και αυτά τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν. Ο Έγινε μία αναφορά στην ελευθερία έκφρασης. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε θέματα που αφορούν την παιδεία. Κάνοντας μία αναδρομή, θα ήθελα να αναφέρω ότι η κυβέρνηση θέλησε να χρησιμοποιήσει την εκπαίδευση σαν έναν τρόπο να ελέγξει την ελευθερία σκέψης. Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ήθελε να προωθήσει ε, αναλυτικά προγράμματα σπουδών εθνικά. Αυτά τα αναλυτικά προγράμματα είχαν στόχο να χρησιμοποιησει την εκπαιδευση σαν εναν τροπο να ελεγξει την ελευθερια σκεψης κανοντας μια αναδρομη στο παρελθον βλεπουμε οτι η κυβερνηση ηθελε να προωθησει αναλυτικα προγραμματα σπουδων εθνικα αυτα τα αναλυτικα προγραμματα ειχαν στοχο να προωθησουν ακολουθήσουν τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας ε, με ένα θετικό τρόπο. Ένα από τα καλά παραδείγματα είναι αυτό. Υπάρχει υλικό το οποίο αναφέρει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έχει βασικό του μέλημα το δημόσιο συμφέρον, είναι ένα προοδευτικό κόμμα, ένα κόμμα που δρά προς το συμφέρον του λαού. Κοιτάζοντας τις απόψεις που εκφράστηκαν σε ό,τι αφορά τα αναλυτικά προγράμματα εθνικής παιδείας, υπάρχουν και ορισμένα άλλα σημεία που θα θέλαμε να αναφέρουμε. Δεν ενθαρρύνθηκαν οι φοιτητές να εκφέρουν μια άποψη προς, προς ε, τις ε, ε, αρχές. Αυτό και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Χονγκ Για τον λόγο αυτό, οι νέοι οργανώθηκαν και στράφηκαν κατά της πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνηση παρόλο το γεγονός ότι ένας από τους αρχηγούς είναι ο Γιούσιν Κέν, η πρόταση που υποβλήθηκε ήταν να αλλάξει το αναλυτικό πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, πρόσφατα οι αρμόδιες αρχές για την εκπαίδευση στο Χονγκ ενδεχομένως σκέφτονται και πάλι να προωθήσουν το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Γιατί εστράφησαν πάρα πολλοί νέοι κατά της κυβέρνησης και ενδεχομένως τα σχολεία είναι υπεύθυνα γι' αυτό. Η κυβέρνηση λοιπόν για μία ακόμα φορά θα επιβάλλει τα δικά της αναλυτικά προγράμματα για να μπορέσει να κάνει, τα λέγαμε, να καθοδηγήσει, να κάνει πλήση εγκεφάλου στους νέους. Στο Χονγκ Κόνγκ, στα, στη δευτεροβάθμια ε, εκπαίδευση υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει σκοπό να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη στους ε, μαθητές. Η κυβέρνηση προτείνει, θέλει να, ε, η πρόταση της είναι, είναι να καταργηθεί το κράτος δικαίου. Λόγω των πρόσφατων συμβάντων στο Χοκόγκ διατυπώθηκαν πάρα πολλές ανησυχίες από πλευράς του πληθυσμού για το κατά πόσον αυτού του είδους τα αναλυτικά προγράμματα καλλιεργούν την κριτική σκέψη των ε, μαθητών. Χρησιμοποιείται επίσης η κυβέρνηση του Πεκίνου για να προωθηθούν αυτοί αυτά τα σχέδια ενώ ορισμένοι πρότειναν τα προγράμματα αυτά να είναι προαιρετικά. Όπως είπαμε, ο στόχος ήταν να προωθηθεί η κριτική σκέψη των ε, μαθητών. Η κυβέρνηση ε, του Χονγκ Κόνγκ προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε για να καταστήλει τα αιτήματα των φοιτητών αλλάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα. Το δεύτερο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο προηγούμενος ομιλητής αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι διαδηλωτές τι προηγούμενες 65 μέρες από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που υπόθηκε ότι η αστυνομία δεν τα κατάφερε να δείξει επαγγελματισμό στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους διαδηλωτές. Αυτό είναι σαφές από τρία σημεία. Οι, χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνει μια αναφορά στις προθέσεις αυτών των κινημάτων. Υπάρχει μία αναφορά ότι κάποιος αστυνομικός έγραψε στη σελίδα του στο facebook ότι οι διαδηλωτές είναι σκουπίδια. Αυτό μας δείχνει ότι στο εσωτερικό των αστυνομικών δυνάμεων στο Χονγκ υπάρχουν ορισμένοι που τρέφουν αρνητικά συναισθήματα για τους διαδηλωτές. Ορισμένοι αστυνομικοί εξέφρασαν σαφώς την άποψή τους ως προς τους διαδηλωτές. Ορισμένοι έβαλαν διακριτικά για να εκφράσουν τις πολιτικές τους πεπιθήσεις πιστεύουν πολλοί ότι οι αστυνομικοί δεν θα πρέπει να έχουν πολιτικές απόψεις που να προωθούν όταν αντιμετωπίζουν τους διαδηλωτές. Το τρίτο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Λό είναι ότι έχουμε στοιχεία που μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο έδρασε ακριβώς η αστυνομία, δημιουργώντας μία χαοτική κατάσταση. Όταν το κίνημα αυτό επεκτάθηκε σε διάφορες περιοχές, οι αστυνομικοί είχαν την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. αντί να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί την κατάσταση με έναν επαγγελματικό τρόπο, άρχισαν τις συλλήψεις των διαδηλωτών. Με αυτόν τον τρόπο κατέστησαν σαφείς τις πολιτικές τους απόψεις. Ο κύριος Λό έκανε μία αναφορά και στο θέμα της λογοκρισίας. Οι κάτοικοι του Χονγκ Κόνγκ ενημερώνονται μόνο από τα μέσα μαζικής ε, ε, ενημέρωσης που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση, είτε πρόκειται για τηλεόραση είτε για εφημερίδες ή ενημερώνονται από τα μέσα εκείνα που προβάλλουν την ιδέα ότι το κίνημα αυτό καταλήψεων οδηγεί σε ένα, σε ένα πολιτικό χάος. Ορισμένες κυβερνητικές εφημερίδες πρόβαλαν και άλλες απόψεις ότι για παράδειγμα ε, πολλά, πολλές πανεπιστημιακές σχολές έχουν ε, λάβει χρήματα από ξένες χώρες, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο χάος στα πανεπιστήμια. Μέχρι στιγμή ε, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε, στις διαδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να, να δώσω εγγυήσεις ότι θα, δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Αυτά είχα να σας πω. ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν θα μείνουν εκεί. Θα μείνουν εκεί, θα συνεχίσουν να ακούνε. Ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν μπορούμε να δώσουμε το λόγο στη Σάρον Ντάμκιν Σόου που είναι μια πολύ γνωστή αγωνίστρια είναι διευθύντρια της οργάνωσης Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κίνα. Και ήδη και σε προηγούμενες εκδηλώσεις έχει παρευρεθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πλέον από, επιπλέον από ε, ακτιβίστρια είναι ειδική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην υπηρετική Κίνα. Να ακούσουμε και εκείνη ε, και μετά θα έχουμε μια συζήτηση και με τους τρεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμβάλλω στην ανταλλαγή απόψεων σε αυτή την κρίσιμη φάση εξελίξεων. Ε, και είναι τιμή για μένα που συμμετέχω με τους δύο άλλους ομιλητές. Έχω μιλήσει στην Επιτροπή σας και στο παρελθόν. Αλλά είναι η πρώτη φορά που μιλάω ως κάτοικος του Χονγκ Κονγκ. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, αλλά με ταπεινοφροσύνη θα σας μιλήσω. Η οργάνωσή μου έχει βάση στο Χονγκ Κονγκ από το 1996 και στην Ευρώπη. Έχουμε εργαστεί για πάνω από 25 χρόνια για να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να υπάρξουν αλλαγές. Ε, μεταξύ αυτών έχουμε υποστηρίξει και τις μητέρες του Tiananmen. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε μέσω του Μηχανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Πρόσφατα, για παράδειγμα, ασχοληθήκαμε με μια επισκόπηση της κατάστασης στην Κίνα και ασχοληθήκαμε και με θέματα ε, εκλογικών δικαιωμάτων. Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ είναι περίπλοκη και ταχαίως μεταβαλλόμενη. Οπότε είναι δύσκολο να έχει κανείς μια έτοιμη ομιλία γιατί από ώρα σε ώρα αυτό το Σαββατοκύριακο ένα κίνημα πολιτικής ανυπακοής ε, που είχε κρατήσει δύο μήνες και που είχε αντιμετωπιστεί με μεγάλο σεβασμό από όλο τον κόσμο, άλλαξε χαρακτήρα, έγιναν βίες εκδηλώσεις και συλλήψεις. Και σήμερα έχει ξεκινήσει από τον Τζόσου Ουάνγκ απεργία πείνας. Και όπως ήδη ακούσατε, οι διοργανωτές της ε, οργάνωσης των καταλήψεων, οι διοργανωτές των καταλήψεων παραδόθηκαν στην αστυνομία. Αντί λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα βασικά θέματα, η κυβέρνηση του Χονγκ Κόνγκ βασίζεται στην ομή βία, ομή αστυνομική βία. Όπως το περιέγραψε ο Δόκτωρ Βάν. Η στάση της αστυνομίας ε, δεν είναι ευσυνείδητη και είναι πολιτικοποιημένη. Επίσης ε, τα δικαστήρια έχουν αξιοποιηθεί για να απελευθερωθούν οι χώροι των καταλήψεων. Η χρήση αυτή των ε, δικαστηρίων για να αντιμετωπιστεί ένα πολιτικό θέμα έχει επικριθεί ως μη κατάλληλη. Και η στάση της κεντρικής κυβέρνησης είναι αυθαίρετη και αυταρχική. Στην υπηρετική Κίνα έχουν εμποδίσει την ενημέρωση για το τι γίνεται. Αυτή τη βδομάδα, αν ψάξει κανείς ε, στο ίντερνετ ε, για το λίμα αστυνομία του Χονγκ Κονγκ δεν θα βρει τίποτα. Έχει λογοκριθεί. Και τα κεντρικά όργανα όπως ε, το πρακτορείο Σιλκουά και η λαϊκή ημερησία τονίζουν ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα διοικηθεί το Χονγκ Κονγκ δεν θα, δεν θα τροποποιηθεί και λένε ότι είναι παρόμοιες εκδηλώσεις που γίνονται στην, ε, στο Χονγκ Κονγκ με τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει στην Ταϊουάν και τη Μέση Ανατολή. Επίσης ε, τονίζουν ότι υπάρχει παρέμβαση ξένων κυβερνήσεων, δυτικών κυβερνήσεων, ότι αυτοί υποδαβλίζουν και χρηματοδοτούν αυτό το κίνημα. Αυτές όμως οι ενέργειες, αυτή η στάση, όχι μόνο καταδεικνύουν ότι αποτυχάνει η κυβέρνηση, δεν μπορούν και να παρεμποδίσουν μακροπρόθεσμα το δημοκρατικό κίνημα. Το δημοκρατικό κίνημα δεν μπορεί πια να σταματήσει. Η αντιμετώπιση του κινήματος είναι πιο δυναμική, πιο δημιουργική και πιο ρευστή. Το κίνημα έχει διατηρήσει ένα θετικό πνεύμα, ακόμη και χιουμοριστικό πνεύμα. Αυτό το βλέπετε. Αυτό το κίνημα ε, ομπρέλα Τώρα λέγεται και κίνημα για shopping. Αυτό είναι η αντιμετώπιση των διαδηλωτών σε αντίδραση ε, στην ε, δήλωση του κυβερνήτη του Βιετνάμ ότι τώρα που ήρθε η κατάληψη σε ένα κεντρικό χώρο αγορών θα πρέπει να πάνε να ψωνίσουν για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία. Ξέρετε ότι παντού στο Χονγκ Κονγκ υπάρχουν ε, τεράστιες οθόνες που δείχνουν ε, ε, διαφημιστικά τρέιλερ για διάφορες ταινίες. Ο κόσμος κάθεται και υψώνει το χέρι κάνοντας το σήμα της δημοκρατίας. Δύο πράγματα μπορούν να ελέγξουν τα αυταρχικά καθεστώτα, την πολιτική ανυπακοή και το χιούμορ. Κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι αυτές οι ενέργειες ε, προκαλούν ριζοσπαστικοποίηση μιας ολόκληρης γενιάς νέων που μεγάλωσαν ζώντας ε, σε καθεστώς ελευθερίας. Η γενιά αυτή είναι τεχνολογικά προηγμένη και μπορεί να δημιουργήσει νέα κοινωνικά μέσα Δικτύωση για να ενημερώσει και να εμπνεύσει τις περαιτέρω εξελίξει. για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και για να συμβάλλουμε επικοδομητικά στην εξέβρεση ειρηνική λύση, είναι σημαντικό να ξεπεράσουμε την πολλωμένη και στατική προσέγγιση των θεμάτων, όπως συζητώνται μεταξύ των ε, διαδηλωτών. Είναι δύσκολη η δημοκρατική διαδικασία, αλλά είναι επίσης συναρπαστική και είναι σε εξέλιξη. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει συνένεση σε διάφορους ε, τομείς, για παράδειγμα. Πρώτον, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο τρόπος ζωής και οι βασικές αξίες του Χονγκ Κόνγκ, κράτος δικαίου, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, όπως έχει ε, όπως ε, υπόσχεται η δήλωση μεταξύ Κίνας και Βρετανίας και ο βασικός νόμος του Χονγκ Κόνγκ. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για τη βιωσιμότητα και σταθερότητα της οικονομίας του Χονγκ Κόνγκ. Δεύτερον, όλοι οι κάτοικοι του Χονγκ Κόνγκ, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, την ηλικία τους και τη θέση τους για το κίνημα καταλήψεων, θεωρούν ότι μόνο μέσω καθολικής ψηφοφορίας μπορεί να προχωρήσουν και καταλαβαίνουν ότι αυτό θα είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. Θα χρειαστούν γενιές. Δεν είναι κάτι που θα επιτευχθεί άμεσα. Να σας μιλήσω για την ε, προσωπική μου εμπειρία. Μίλησα με ταξιτζίδες, με πλανόδιους πολιτές και όλοι συμφωνούν. Μίλησα ακόμη και με νέα παιδιά και με τους ε, γονείς τους που μοίραζαν αυτές τις κίτρινες κορδέλες και που είναι το σύμβολο Ρώτησα λοιπόν τους γονείς, καταλαβαίνουν τι κάνουν. Και οι γονείς μου είπαν, ρωτήστε τα παιδιά. Ρώτησα ένα αγοράκι που είπε, είμαι πέντε ετών. Πέντε είπα, και τι ακριβώς κάνεις. Και μου απάντησε, χωρίς να διστάσει, θέλω να υπάρξει καθολική ψηφοφορία. Και το κοριτσάκι είπε, είμαι έξω ε, γράφω, όχι, συγγνώμη, είμαι πέντε χρόνια και ξέρω να γράφω. Και τι μπορείς να γράψεις, είπε. Θέλω ε, κάθε πολίτης να έχει ε, ψήφο, είπε και το κοριτσάκι. Και ξεπλάγει. Και είπα στη μητέρα τους, μα είναι πέντε ετών. Και η μητέρα μου είπε ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους φοιτητέ, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε και την επόμενη γενιά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ειρηνική και βιώσιμη λύση ε, στον αγώνα για δημοκρατία και εκλογικά δικαιώματα των κατοίκων του Χονγκ Και αυτά θα έχουν επιπτώσεις και στην υπηρετική Κίνα. Αυτό φαίνεται από το γεγονό ότι έχει ε, επιβληθεί λογοκρισία και έχουν συλληφθεί πάνω από 100 Κινέζοι από την υπηρετική Κίνα που υποστηρίζουν την, ε, τις καταλήψεις στο Χογκόν και θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις και στην ευρύτερη περιοχή. Και φυσικά δεν καθησυχάζουν καθόλου τους κατοίκους ε, της Ταϊουάν ότι αν ε, ενωθούν με την Κίνα θα έχουν διαφορετικό σύστημα. Δεν θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσει ότι είναι εσωτερικό θέμα του Hong ε, της Κίνας συγγνώμη, τα θέματα αυτά. Αυτά τα είπαν και στη Βρετανική Βουλή χθες και επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε πρόσβαση στο Χονγκ για να γίνει μια έρευνα. Και είναι σαφές ότι όλοι οι κοινοβουλευτικοί πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στο Χονγκ Κόνγκ και έχουν και ρόλο για να διασφαλίσουν ότι η κοινή δήλωση αυτή μεταξύ Βρετανίας και Κίνας και η υποσχέση που περιείχε πρέπει να τηρηθεί. Οποιαδήποτε άλλη στάση θα ήταν ανεύθυνη. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω, όπως και οι Βρετανοί κοινοβουλευτικοί, να καταλάβετε ότι έχετε σημαντικό ρόλο να παίξετε. Θεωρώ λοιπόν ότι με, με βάση το άρθρο 21 της συνθήκης χρειάζεται συνέπεια στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης και ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή θα καθοδηγούνται από τις αρχές που έχουν εμπνεύσει την ίδρυσή της, την εξέλιξή της, τη διεύρυνσή της και προσπαθεί να προωθήσει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την καθολικότητα και το αδιέρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την αλληλεγγύη. Όσο λοιπόν προσπαθεί η Ένωση να ακολουθήσει και να σεβαστεί αυτή την πολιτική σε όλους τους τομείς της διεθνούς πολιτικής, σε σχέση με το Χονγκ θα ήθελα να σας πω ότι ναι μεν είναι σημαντικός εταίρος σας η Κίνα και το Χονγκ Κόνγκ και γι' αυτό μια κυβέρνηση που δεν λογοδοτεί στο λαό της, που δεν δρά διαφανώς, που δεν τηρεί τις υποσχέσεις της, δεν θα είναι καλός εμπορικός εταίρος. Ο διάλογος ε, Ένωσης Κίνας ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα λάβει χώρο 8 και 9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Ως οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών έχουμε ε, πλήρη αντίληψη του πόσο δύσκολες είναι αυτές οι συζητήσεις, οι διμερείς. Και από ό,τι καταλάβαμε το Χονγκ Κόνγκ δεν θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό διότι θα συζητηθούν θέματα όπως η ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα ε, και στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου ενημέρωσης. Θα πρότεινα λοιπόν η ενωσιακή αντιπροσωπεία σε αυτό το διάλογο να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς την κινέζικη κυβέρνηση <clears throat> για τη σημασία επαφής με τους ηγέτες αυτού του κινήματος, επαφής με το λαό του Χονγκ να υπάρξει επικοδομητική πρόοδος. Υπενθυμίζουμε ότι ο ειδικό αντιπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ένωσης, κύριος Λαμπρινίδης, επισκέφθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 την Κίνα και ήταν επικοδομητική η επίσκεψή του. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να δούμε μια παρόμοια πρωτοβουλία του για να υποστηρίξει τον αγώνα του λαού του Χονγκ Επιπλέον, Να θυμηθούμε, δεν είναι η πρώτη φορά που ενωμένα οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ αντιστάθηκαν στις προσπάθειες περιορισμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Το Χονγκ Κονγκ είναι το μόνο μέρος στην Κίνα τα τελευταία 25 χρόνια όπου πάνω από 100.000 άτομα έχουν συγκεντρώνονται κάθε Τετάρτη Ιουνίου επέτειο της, εξε, καταστολής στο Τιέναν στην, ε, στους κήπους ε, της Βικτόρια. Επίσης έχουν εντεθεί σε ένα νόμο για την ασφάλεια και το άρθρο 23 αυτού του νόμου που θα έδινε τη δυνατότητα στην ε, κυβέρνηση του Χονγκ να καταπνίξει την ελευθερία έκφρασης. Αυτή η ενότητα νέων ηλικιωμένων ε, ηγετών ε, του επιχειρηματικού κόσμου, πανεπιστημιακών και τέτοια, μόνο η κοινή αυτή δράση οδήγησε στην απόσυρση αυτού του νόμου και στην παρέτηση αυτού που τον είχε προτείνει. Και πρόσφατα ένας 16χρονος οργάνωσε μία, ε, ίδρυσε μία οργάνωση που έχει ε, οργανώσει πολλές εκδηλώσεις, συζητήσεις, διαδηλώσεις όπου εκφράζονται ανοιχτά κατά κάθε προσπάθειας λογοκρισίας. Έχουν συλλέξει πάνω από 100.000 υπογραφές και ο Τζο Σουάν, είναι ο κεφαλής αυτής της οργάνωσης δήλωσε ότι η οργάνωσή του γράφει ιστορία και θεωρεί ότι θα υπάρξει σύντομα ένα θαύμα. Είχε δίκιο. Όταν το ρώτησαν ε, τι διδάγματα έχει εξαγάγει, απάντησε ότι πρέπει να εμείνουμε. Ο καθένας μας μπορεί να είναι πραγματικά πολίτης. Η πρόκληση για όλους μας είναι πώς θα τους στηρίξουμε, πώς θα διασφαλίσουμε ότι το τίμημα που ε, θα χρειαστεί να ε, πληρώσουν δεν θα το φέρουμε βάρος στη συνείδησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο έχω ζητήσει τον λόγο. Πρώτος ο Γιολάινεν. Παρακαλώ είναι υπεύθυνο αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τη σχέση με τη λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα. Και μετά ο κύριο Παντσέρη. Και μετά ο κύριο Τόκιο. Ο κύριο Λάινεν, λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, ακούνε οι ε, φίλοι μα στο Χονγκ Κονγκ. Είναι καλύτερα να μιλήσω αγγλικά. Μα ακούτε στο Χονγκ Κονγκ. Έχετε διερμηνία. Α, πολύ ωραία. ωραία. Άρα μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και από το Χονγκ Κόνγκ. Θαυμάσια τεχνολογική βοήθεια μας επιτρέπει να επικοινωνούμε παρά την απόσταση. Όπως είπατε και εσείς εδώ στο Προεδρείο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τελευταία του Ολομέλεια συζήτησε το θέμα του Χονγκ Κόνγκ, έγινε μια πολύ έντονη συζήτηση για το φοιτητικό κίνημα, για το, κίνημα, για το κοινωνικό κίνημα, το κίνημα της κοινωνίας των πολιτών. Και σήμερα εδώ, ως Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνεχίζουμε τη συζήτηση όπως βλέπετε. Βλέπετε λοιπόν ότι παρακολουθούμε πολύ στενά αυτά που συμβαίνουν στο Χονγκ Κόνγκ και οπωσδήποτε υπάρχει πολύ μεγάλη συμπαράσταση του Κοινοβουλίου στον αγώνα σας για δημοκρατία και ελευθερία. Αυτό είναι στο γονιδίωμα του Κοινοβουλίου. Είμαστε υπέρ της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε λοιπόν. Μας είπατε ότι η διαδικασία εκδημοκρατισμού δεν μπορεί πλέον να σταματήσει. Και ακούσαμε επίσης όμως ότι στο Χονγκ Κόνγκ αυτή τη στιγμή περιορίζονται τα δημοκρατικά δικαιώματα. Προς ποια κατεύθυνση λοιπόν πάει, ποιος θα, ε, ποιος θα έχει το πάνω χέρι, το κίνημα ή οι αρχές. Και η στρατηγική του κινήματος διαμαρτυρίας ε, ξεκινήσατε με διαδηλώσεις, ε, με καταλήψεις οδών. Βέβαια αυτό έχει κάποιους περιορισμούς γιατί κάποτε ο πληθυσμός θέλει επίσης να μπορούν να κινηθούν τα αυτοκίνητα και οι πολίτες. Ξέρουμε ότι αυτά τα κοινωνικά κινήματα μπορεί να αναπτυχθούν και μετά ε, τίθεται το ερώτημα τώρα τι θα κάνουμε. Θα υπάρξει ριζοσπαστικοποίηση, προς ποια κατεύθυνση θα πάμε. Και εκεί μπορεί να προκύψουν διασπάσεις. Κάποιοι που θέλουν πιο ριζοσπαστικές μορφές πάλι, ενώ οι άλλοι ψάχνουν νέες μορφές πάλι, ε, να γίνει το κίνημα ε, με τις ομπρέλες, κίνημα για ψώνια κτλ βλέπουμε διάφορες μορφές έκφρασης. Για μένα είναι σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρξει βία. Δεν θα επιτύχει τίποτα η βία. Μόνο μέσω πολιτικής δράσης. Πρέπει να ψάξουμε πολιτικές μορφές πάλι. Κοιτάξτε, Πιστεύω Πιστεύουμε ότι είναι θέμα της κυβέρνησης του Πεκίνου. Σας απαντάει κύριε, σας απαντάνε κύριε Λάινα. Παρακαλώ, ε, συνεχίστε κύριε Λάινα. Έχετε δύο λεπτά, όχι. Μάλλον έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει, αλλά ξέρω ποιος θα χάσει. Χάνουν οι κυβερνήσεις του Μπέιτζινγκ και του Hong Κονγκ για τα επόμενα χρόνια εάν δεν βελτιώσουν την κατάσταση της δημοκρατίας του Χονγκ Κονγκ, θα έχουν μεγάλες δυσχέρειες. Δεν θα μπορούν να κυβερνήσουν ουσιαστικά το Hong Kong. Και αυτό οπωσδήποτε θα αποτρέψει και την Ταϊβάν από περαιτέρω συνεργασία με την Κίνα. Δηλαδή από πλευρά ε, ενδεχομένη ε, επανενοποίησης Ταϊβάν ε, υπηρετική Κίνας. Οπωσδήποτε βεβαίω θα χάσει την εμπιστοσύνη η κυβέρνηση του Χονγκ την εμπιστοσύνη του λαού. Κοιτάξτε, η αστυνομία μας είχε υποσχεθεί ότι δεν θα παρεμποδίσει τις δραστηριότητες επιτήρησής μας. Και τώρα δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και μας περιορίζουν. Ελπίζουμε να μπορέσετε να μας βοηθήσετε, να μας ε, χορηγήσετε προστασία. Για να μπορούμε να ε, παρακολουθούμε εάν γίνονται παραβιάσεις των δικαιωμάτων μας στο έδαφος ε, δηλαδή επιτόπου. Και ε, επίσης να προωθήσετε το δικαίωμα καθολικής ψηφοφορίας. Δεν είναι δυνατόν ε, η Κίνα να αρνείται τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Έχουν δεσμευτεί μέσω διεθνών συμβάσεων να εφαρμόσουν το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας. Κύριε Λάου, κύριε Λάου, κύριε Λάου, να ακούσουμε τον κύριο Λάινεν. Και κοιτάξτε, υπάρχουν διεθνές προδιαγραφές. Ευχαριστώ κύριε Λάου. Συνεχίστε κύριε Λάινεν. Μα τελείωνα, τελείωνα. Έχουμε τον ε, διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ένωση Κίνα και σας διαβεβαιώ ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πάει στην Κίνα το Μάρτιο θα επισκεφθεί και το Χονγκ Κονγκ και θα έχουμε τότε την ευκαιρία να σας ε, συναντήσουμε και να συνεχίσουμε το διάλογο που ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάιναν. Ο κύριος Παντσέρη. Εγώ θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις και να εκφράσω ορισμένες σκέψεις, ελπίζοντας να τύχω μια απάντησης. Όπως διαβάσαμε χθε το απόγευμα, οι τρεις ειδητέ της ομάδας Occupy Hong Kong εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να παραδοθούν στην αστυνομία αναγνωρίζοντας ότι είχαν διαπράξει κάποια εγκληματική πράξη. Ζητώντα από τους διαδηλωτέ να αποσυρθούν. Δεν ξέρω εάν όντω είναι έτσι τα πράγματα, να αυτό συνέβη από μια αστυνομία που, η οποία δεν έχει πλέον κανέναν έλεγχο στι πράξεις της ή αν έχει σχέση με αυτό το κίνημα κατάληψης των δρόμων και των πλατιών. Η δική μου προσωπική άποψη και η αίσθηση που έχω, πέρα βεβαίως από την απεργία πείνας, είναι ότι υπάρχουν πολλοί φοιτητέ οι οποίοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να αποχωρήσουν και υπάρχει ο κίνδυνος ότι αυτή η κινητοποίηση θα μπορούσε να εξαντληθεί με την παρακάτω αντίφαση. Από τη μία πλευρά κίνησε ιδιαίτερα την προσοχή όλων των διεθνών μέσων, εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήραμε ορισμένε πρωτοβουλίε και από την άλλη πλευρά αποτελέσματα τα οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος για περισσότερη δημοκρατία και για άμεση καθολική ψηφοφορία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα ε, περισσότερο ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά κυρίως την Κίνα και όπως αναφέρθηκε θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του άρθρου 21 της Συνθήκης Λισαβόνας. Μετά από αυτή την ακρόαση θα μιλήσουμε για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα θίξουμε και το θέμα της συνοχής των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν. Κατά κάποιον τρόπο θα θέλαμε να καταλάβουμε αν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τρεις στόχους. Πρώτον, να εδρεωθεί μια πιο σωστή σχέση συνεργασίας με την Κίνα. Δεύτερον, το να μην θεωρείται το Χονγκ σαν ε, ε, ένα σκόμπος χρηματοπιστωτικό, αλλά μια πραγματικότητα ε, που αφορά μεταξύ των άλλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να κινηθούμε σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε ουσιαστικά στις κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις που ακόμα λαμβάνουν χώρα στο Χονγκ Κόγκ. Ο κύριος Παντσέρη είναι ο συντάκτης της έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα δούμε μετά. Δηλαδή ε, συμμετέχει άμεσα στην προσπάθεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Τόκες. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Διαβάζω σε αυτό το έγγραφο που λάβαμε σήμερα ότι, ότι το καθεστώς της Κίνας έχει μη δημοκρατικό χαρακτήρα. Ε, είναι κάπως ε, εφημισμός αυτή η διατύπωση. Ε, αν θυμάστε, το 1999 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε τις δύο απολυταρχικές ε, ολοκληρωτικές μορφές διακυβέρνησης και τον κομμουνισμό και τον εθνικό σοσιαλισμό. Η Κίνα είναι κομμουνιστικό κράτος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι σαφές ότι ο κομμουνισμός ναι μεν κατέρευσε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη στη Ρουμανία είναι σήμερα επέτειος της, κατα... της του πριν από 25 χρόνια όμως στην Κίνα και στην Κούβα εξακολουθεί να υπάρχει κομμουνισμός και πρέπει αυτό να το καταγγείλουμε και να το καταπολεμήσουμε δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε ο κομμουνισμός να καταλάβει και το Χονγκ Κόνγκ. Όταν υπογράφηκε η συνθήκη για την παράδοση της, ε, του Χονγκ Κόνγκ στην Κίνα, η αρχή ήταν μία χώρα, δύο συστήματα. Μόνο έτσι συμφωνήθηκε να παραχωρηθεί το Χονγκ Κόνγκ στην Κίνα. Πρέπει να επιμείνουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η αρχή. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταγγείλει τον κομμουνισμό. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει πρόβλημα και με τους Ουιγούρους στην ε, Δυτική Κίνα. Ξέρουμε το πρόβλημα που υπάρχει και στο Θιβέτ. Θα κάνουμε μια κρόση για τα θέματα αυτά σήμερα. Πρέπει οπωσδήποτε, εφόσον εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως υποεπιτροπή, να ασχοληθούμε με αυτά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Βαλεντιάνο που οργάνωσε αυτήν την ακρόαση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα θέματα αυτά να είναι μονίμως στην ημέρηση διάταξη. Η κατάσταση του Χονγκ Κόνγκ πρέπει να μας απασχολήσει. Και κάτι ακόμη. Η Κίνα λέει ότι δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές ε, υποθέσεις της ε, Κίνας. Και ο Τσαουσέσκου πριν από 25 χρόνια έλεγε ότι κανείς δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της ε, Ρουμανίας. Τα έχουμε ξανακούσει λοιπόν αυτά και δεν είναι δυνατόν να τα δεχτούμε. Ευχαριστώ πολύ γιατί πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριος ε, Τζισεβίτσιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, τους ε, συνδιαλεγόμενούς μας που βρίσκονται πάρα πολύ μακριά για το μήνυμα που μας ε, ε, απέστειλαν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη της έκθεσης ε, του κυρίου Παντσέρη την οποία θα συζητήσουμε και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πρέπει να καταλαβαίνουμε καλύτερα εμείς ως μέλη της Επιτροπής αυτής ε, ο όλο ένα και αυξανόμενος ε, ε, ρόλος της Κίνας και η οικονομική της ανάπτυξη θα έπρεπε να συνάδει με δεσμεύσεις για τις πολιτικές ελευθερίες. Αν θέλει λοιπόν η Κίνα να έχει σημαντικότερο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία πρέπει να καταλάβει ε, ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος ε, για τα ε, θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό το μήνυμα πρέπει να αποστέλλεται από όλους εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση ε, στους εκπροσώπους του Χονγκ Κονγκ. Ε, η ανταπόκριση άλλων μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Υπάρχει, υπήρξε επαφή με άλλους αντιφρονούντες ή με άλλους ε, με άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που δραστηριοποιούνται τοπικά στο Χονγκ Κόνγκ και ποιες είναι οι προσδοκίες των ε, εκπροσώπων του Χονγκ Κόνγκ από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς ε, να σας υπενθυμίσω ότι η ομάδα του ΕΛΚ έχει υποστηρίξει τη συζήτηση αυτή, τον εγγραφή δηλαδή στην ημερήσια διάταξη. Ε, εγώ ε, θα ήθελα να είναι κατεπήγον, αλλά ήταν νομίζω καλό το ότι μπορέσαμε να το συζητήσουμε και στο Στρασβούργο μου κάνει εντύπωση ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας ε, δεν συμπεριλαμβάνει το θέμα του Χονγκ Κόνγκ. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Λαμπρινίδης πρέπει να μεταβεί στο Χονγκ Κόνγκ το συντομότερο δυνατό. Νομίζω ότι είναι μια ελάχιστη χειρονομία η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται όχι μόνο από συνοχή αλλά και από ταχύτητα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσουν οι εξελίξεις, ούτε μπορούμε να αναβάλουμε ε, την ε, συμμετοχή μας. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Τόκιος προηγουμένως, θα ήθελα να πω ότι η ιδέα μία χώρα, δύο συστήματα είναι μία αυταπάτη. Η μοναδική πραγματικότητα που βλέπουμε να ισχύει, ε, που, που βλέπουμε ότι πρέπει να ε, ισχύσει, είναι ο εκδημοκρατισμός της Κίνας. Πιστεύω ότι πραγματικά Αυταπατώμεθα αν πιστεύουμε ότι μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο στο μέλλον η ιδέα μία χώρα, δύο συστήματα. Η μόνη πραγματική και βιώσιμη λύση είναι ο εκδημοκρατισμό τη Κίνα και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποστείλει αυτό το μήνυμα σαφέστατα και χωρί κανέναν απολύτω δισταγμό. Και όπως είπε και κάποιο από του προσκεκλημένου μα, δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιο σοβαρό εμπορικό εταίρος αν αυτός ε, ο εταίρος δεν ε, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, να δώσω το λόγο στους ε, εμπειρογνώμονές μας από το Χονγκ Κόνγκ. Δύο λεπτά παρακαλώ και μετά και στην κυρία Κονγκ. Παρακαλώ έχετε το λόγο. συμφωνώ ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα μηνύματα ε, για το κίνημα του Χονγκ Κόνγκ να περάσουν στην επιρροτική Κίνα γιατί υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα και πολλές διαφωνίες. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες που έρχονται στο Χονγκ Κόνγκ και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την κατάσταση του Χονγκ Κόνγκ η κινέζικη προπαγάνδα κατά το ε, Hong και κατά του Hong Kong και του κινήματος αυτούς δεν βοηθά τον κόσμο να καταλάβει την κατάσταση ε, στο Hong Kong. Ούτε και το έγγραφο αυτό το οποίο λάβατε Όσον αφορά τώρα κατά πόσο υπάρχει, ε, ε, υπάρχουν υποστηρικτές του κινήματος στην Κίνα, ακόμη και να υπάρχουν, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για αυτούς τους ε, ανθρώπους. Και όσον αφορά, για το θέμα, όσον αφορά το θέμα του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Χονγκ Κόνγκ. Αυτή τη στιγμή η φόρμουλα είναι η εξή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών ε, ε, στο Χονγκ Κόνγκ βάσει του ε, βασικού νόμου, του μήνυ συντάγματος. Όμως γίνεται αυθαίρετη ερμηνεία αυτού του νόμου από την Κίνα, από τις κινέζικες αρχές. Οπότε... Πρέπει να ε, λέτε ε, ότι πρέπει να ερμηνεύετε ε, συμφώνος προς το ε, Διεθνές Σύμφωνο για τα πολιτικά ε, δικαιώματα. Ο βασικός νόμος πρέπει βάσει διεθνών προτύπων να ερμηνεύεται. Η Κίνα έχει αρχίσει τώρα να αρνείται τη χρήση της κοινή δήλωσης, της, της συνοβρετανικής δήλωσης και αυτό πραγματικά αποτελεί μια ε, ε, κατάφορη ε, άρνηση διεθνών δεσμεύσεών τους. Δεν, δεν, δεν σέβονται πια και δεν αναγνωρίζουν συνθήκες. Αν δεν αντισταθείτε σε αυτό θα είναι πραγματικά τρομερό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ εσείς. Σε σχέση με τα στοιχεία ε, που άκουσα, όταν μιλάτε για το θέμα της μίας χώρας δύο συστημάτων και λέτε ότι είναι αυταπάτη και ότι είναι ε, ο εκδημοκρατισμός της Κίνας που είναι η μοναδική βιώσιμη λύση, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ε, στο δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων της πολιτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του Χονγκ Κόνγκ που θα αρχίσει κατά πάσα πιθανότητα τον Ιανουάριο του 2015. Αλλά για την ώρα δεν έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία ε, της έναρξης του δεύτερου γύρου των διαβουλεύσεων. Φοβούμε όμως ότι αν δούμε τον πρώτο γύρο των ε, ε διαβουλεύσεων, Υπήρξαν μόνο οι κυβερνητικές απόψεις και οι συντηρητικές απόψεις που ακούστηκαν σε σχέση με τα ρύθμιση. Κατά τη διάρκεια της ε, διαβούλευσης ε, υπήρξε ένας αξιωματούχος ε, της Κίνας Ο Κινέζος εκπρόσωπος λοιπόν στο Χονγκ Κόνγκ λέει συνεχώς ότι δεν πρέπει να ε, ε, υπάρχει διαφωνία ε, ως προς το διορισμό των υποψηφίων από, το, από την Κίνα και ότι έχουν στο μυαλό τους το καλύτερο συμφέρον του Χονγκ κλπ. Αυτό έγινε στον πρώτο γύρο των διαβουλεύσεων και είναι αυτό που θα συμβεί και στο δεύτερο γύρο των διαβουλεύσεων κατά πάσα πιθανότητα. Κάτι ακόμη Συνεχώς λοιπόν ε, οι εκπρόσωποι της Κίνας ε, αναφέρουν ότι το μόνο που θέλει το Χονγκ Κόνγκ είναι άμεση καθολική ψηφοφορία. Ε, για, το γνωρίζουμε ε, ότι άμεση καθολική ψηφοφορία, αλλά όχι δημοκρατία, είχε και η ναζιστική Γερμανία και η Βόρεια Κορέα. Αυτό δεν αρκεί και ουσιαστικά αυτή είναι μια προπαγάνδα που προωθεί η Κίνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η άμεση καθολική ψηφοφορία λύνει τα προβλήματα της δημοκρατίας. Αν υπάρχουν τέτοιου είδους αρνητικές ή παραπλανητικές πληροφορίες, ε, ουσιαστικά θα αποδυναμωθεί η διαδικασία του εκδημοκρατισμού. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά η κυρία Σάρον Τάνκισουν. Και μετά θα δώσω το λόγο στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για τα όσα σημαντικά θέματα έφτιαξαν και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα όσα συγκεκριμένα ακούσαμε σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες συστάσεις αλλά και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Θα ήθελα εν συντομία, γιατί δεν έχουμε χρόνο, σχετικά με το θέμα ποιος θα είναι ο νικητής και ποια θα είναι η στρατηγική καταρχάς βρίσκεται στο DNA του Κομμουνιστικού Κόμματος να είναι, της Κίνας να είναι αντιδημοκρατικό. Είναι στο DNA τους η ανάγκη διατήρηση του ελέγχου. Συνεπώς ε, θα συνθλιβεί οποιαδήποτε προσπάθεια εδραίωσης μιας πολιτιστικής ταυτότητας το κράτος δικαίου. Μιλώντας πάντοτε για το DNA, το κράτος δικαίου δεν είναι στην Κίνα αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος. Ε, ε, ε, δεν μιλάμε για κράτος δικαίου, μιλάμε για μια διακυβέρνηση με νόμους. Αυτή είναι μια ε, διάκριση που θα πρέπει να γίνει και για να μπορέσει να υπάρξει εκδημοκρατισμός και στην υπόλοιπη Κίνα θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες ε, βάσει των οποίων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους, να συμμορφώνονται με τον ε, νόμο και το ίδιο το κόμμα. Αυτό είναι κάτι που αναφέρθηκε στα συμπεράσματα της Επιτροπής τον προηγούμενο μήνα. Δεν έγινε μια άμεση αναφορά στην ε, ανταλλαγή απόψεων με την κινέζικη αντιπροσωπεία έγινε αναφορά στις ε, πολιτικές ε, ε, επιτροπές που είναι εξάρτητες από τη δικαιοσύνη. τελικά συμπεράσματα η Επιτροπή είπε ότι θα ήθελα να δοθεί επιτροπή στα μέτρα που θα υιοθετηθούν για να αντιμετωπιστεί το σύστημα των παρεμβάσεων στην δικαιοσύνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την ανησυχία μας για όσα συμβαίνουν. Υπάρχουν νέα κινήματα των πολιτών και στην υπόλοιπη Κίνα σε μια προσπάθεια συμμετοχής, για μια προσπάθεια για να υπάρξει η μεγαλύτερη ανεξαρτησία, για μια διεθνή συμμετοχή. Αυτό ε, δεν γίνεται δεκτό, οι άνθρωποι αυτοί έχουν φυλακιστεί για τις πράξεις τους και μόνο. Αυτό που δεν κατάφεραν να ελέγξουν είναι την διαδικτυακή ε, σύνδεση. Υπάρχουν δραστηριότητες των πολιτών στο διαδίκτυο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. άλλο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το Hong και η πόλη Κίνα καταβάλουν προσπάθειες για μία χώρα ένα σύστημα, αλλά βεβαίως υπάρχει θέμα ανθρώπων και επενδύσεων. 7 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο, ο πληθυσμός ε, είναι 7 εκατομμύρια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Κινέζοι που έρχονται για να σπουδάσουν ή για να κάνουν διακοπές ή έρχονται για επιχειρηματικέ δραστηριότητες στο Χονγκ Μπορείτε να φανταστείτε τι συνεπάγεται αυτό. Το εδώ είναι μια ιστορία σκύλου που κυνηγάει την ουρά του και, αυτό, ε, και σε αυτό είναι θεατής ε, το Πεκίνο. Βλέπετε πως ε, οι Κινέζοι παροτρύνουν το Χονγκ Αυτό είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση. Αυτό δεν γίνεται με έναν τρόπο επίσημο γιατί θα ήταν επικίνδυνο, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει στήριξη ιδιαίτερα διαδικτυακά και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ε, προστατεύσουμε υπό το ε, κάλυμα της ελευθερίας του συναθρίζεστε και της ελευθερίας ε, της, του λόγου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έλλης Μάθιος που είναι επικεφαλής τμήματος στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ και καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να πάρουμε το λόγο στο τέλος ε, αυτής ε, της ε, συζήτησης. Παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυ στο Χονγκ Κόνγκ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και νομίζουμε ότι υπάρχει ένα διακύβευμα εδώ στο μέλλον του Χονγκ Κόνγκ. Παραμένει βεβαίως, παραμένουν τα πράγματα καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστούν και θα πρέπει να σκεφτούμε τα τόσα συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα και ζητάμε από όλους να ξεκινήσουν ένα διάλογο σε μια προσπάθεια ανέβρεσης μιας επικοδομητικής λύσης. Αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια του βασικού δικαίου και του συνάγματος του Χονγκ Κόνγκ. Βεβαίως και οι δύο πλευρές ε, θα πρέπει να τα συνυπολογίσουν όλα αυτά. Ε, το Χονγκ έχει καθοριστικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω θέλουμε να υπάρχει κράτο δικαίου, ελευθερία τη έκφραση. Υπάρχουν και πάρα πολλέ οικονομικέ σχέσει. Είναι βασικό εμπορικό μα ε, εταίρο και έχει στενέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Επτά δεσμευτήκαμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύσαμε, δημοσιεύουμε οι οικονομικές εκθέσει, τις οικονομικές ε, γεωπολιτικές εξελίξεις ε, στο Χονγκ από τότε που πέρασε στην ε, Κίνα. Είναι πάρα πολύ σημαντική για μας είναι σημαντικές δημοκρατικές εξελίξεις η σταθερότητα στο Χονγκ Κονγκ. Βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται από το σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων ε, ελευθεριών στο Χονγκ από το σεβασμό του δικαιώματος ε, του συναθρίζεστε, το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και σε ένα ανεξάρτητο βεβαίως δικαστικό σύστημα. να αναφέραμε ότι υποστηρίζουμε την ε, εκλογή της, την καθολική ψηφοφορία. Αυτά είναι όλα θέματα που έδειξαν και ε, οι ομιλητές πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση η οποία λογοδοτεί, συμβάλλει σε όλα αυτά και με, ε, με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την αξιοπιστία της. Όλα λοιπόν αυτά τα θέματα συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Καταλαβαίνουμε ότι η απόφαση που υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο της Κίνας απογοήτευσε πολλούς στο Χονγκ γιατί ήταν μια στενόμυαλη απόφαση και αυτό αποτέλεσε την απαρχή των διαδηλώσεων. Εμείς ε, μεταφέραμε ε, τις ανησυχίες μας και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι συχνά θέτουμε το θέμα αυτό στους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών στο Κονγκ Κονγκ και με τις, τις κινέζικες ε, ε αρχές υπάρχει, έχουμε, εκπροσωπούμεθα στο Χονγκ Κονγκ, υπάρχει αντιπροσωπεία και ε, υπάρχει συνεχής ενημέρωση, συνεχής ε, αναφορά και κυρίως τις τελευταίες ε, δύο εβδομάδες. Βεβαίως υπάρχει και συντονισμός με τις χώρες μέλη εδώ στις Βρυξέλλες, χώρες μέλη που εκφράζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα μέχρι Τώρα οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικέ μέχρι στιγμή βέβαια. Είναι σαφές για μας ότι υπάρχει ελαστικότητα για να βρεθεί μια λύση συμβιβασμού στα πλαίσια της απόφασης του NPCSC e και βεβαίως υπάρχει μια κλιμάκωση από πλευράς ε, της αστυνομίας, κάτι ιδιαίτερα ε, ατυχές θα ήθελα να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπαμε σε μια προσπάθεια περιορισμού και από τις δύο πλευρές. Πιστεύουμε ότι είναι λυπηρό ότι σταμάτησαν οι συνομιλίες με τους φοιτητέ και διαβουλευσει και πάλι καθυστέρησαν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει και πάλι να ξεκινήσει ο διάλογος και θα επιθυμούσαμε να καταβληθούν προσπάθειες για ένα πιο δίκαιο ε, εκλογικό σύστημα που θα επιτρέψει μεγαλύτερη συμμετοχή των κατοίκων του Χονγκ Κόνγκ. Υπάρχει μια εδρεωμένη σχέση με τις αρχέ του Χονγκ Κόνγκ. Διεξάγεται διάλογο σε αιτήσια βάση. Από πλευρά μας υπάρχει να παράσχουμε βοήθεια και να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές εξελίξεις και θα θέλαμε να τονίσουμε ότι συμφωνούμε με τα όσα είπαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του Χονγκ Κονγκ και προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα, τελειώνοντας την παρέμβασή μου, να αναφερθώ στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον οποίο έγινε αναφορά, βεβαίως θα μπορούσα να πω ότι επειδή υπάρχουν βασικές ανησυχίες όχι μόνο στο Χονγκ Κόνγκ αλλά και στην Κίνα μας ε, βοηθά να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντική είναι η κατάσταση. Βεβαίως θέλουμε να επιτευχθεί η ε, ελευθερία του συναντρίζεστη, η ελευθερία της έκφρασης, η καθολική ψυχοφορία και βεβαίως αυτά είναι δικαιώματα που θα τεθούν για μία ακόμα φορά στο διάλογο για τα ανθρωπιστικά θέματα. Πριν καταλήξουμε, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μας ε, στο Χονγκ Κόνγκ και την ε, ειδικό εδώ στο πλάι μου για τη συμμετοχή τους. Αυτά που θέλω να πω μετά την παρέμβαση του κύριου Έλλης είναι ότι συνέβη κάτι καινούριο, πιστεύω. Κάτι καινούριο στο Χονγκ και ίσως, ίσως, επειδή συμβαίνουν ε, διαφορετικά γεγονότα, διαφορετικού τύπου, θα πρέπει και η Ένωση να τροποποιήσει τη στάση της. Δεν μπορεί να κάνουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στις σχέσεις, στις σχέσεις μας με την Κίνα. Και στην υπηρετική Κίνα, αλλά κυρίως στο Χονγκ Υπάρχει πραγματική πίεση από τους διαδηλωτές. Ακούσαμε τους προσκεκλημένους μας. Μας εξήγησαν ε, ε, ποια είναι η στάση της αστυνομίας και κανείς δεν αφισβήτησε αυτά που είπαν. Και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το Χονγκ δεν είναι απλώς ένας ενδιαφέρον εμπορικός εταίρος. Έχουμε λοιπόν διάλογο με την Κίνα. Το Χονγκ Κονγκ πρέπει να είναι στοιχείο κλειδί στο διάλογο αυτό, όχι απλώς ένα στοιχείο μεταξύ άλλων. Τι εννοώ. Συμβαίνει κάτι και η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλώς πρέπει να το λάβει υπόψη της, αλλά πρέπει να βοηθήσει για να προχωρήσουμε στον εκδημοκρατισμό όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Οπότε πρέπει να σας πω ότι περίμενα κάτι περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τη στάση της για το Χονγκ Κόνγκ. Ιδίως όταν έχουμε ενώπιόν μας ε, αγωνιστές, άτομα που κάνουν μια εργασία πολύ σοβαρή και που ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν Οπότε από την ε, πλευρά μου και από την πλευρά της Επιτροπής μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε το θέμα της ενίσχυσης ε, του εκδημοκρατισμού, της πορείας εκδημοκρατισμού του Χονγκ Κόνγκ να μείνει στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο για την κοινωνία του Χονγκ Κόνγκ, αλλά και για την κοινωνία της Κίνας, γενικότερα, για όλους μας για όλους όσους πιστεύουμε στη δημοκρατία για όλους ανεξάρτητα από που βρίσκονται, ανεξάρτητα από την πολιτική τους πραγματικότητα. Γι' αυτό δουλεύει η Επιτροπή μας. Χάρη στην ε, αποφασιστικότητά μας, στη στήριξή μας, στα πλαίσια του διαλόγου, του πολιτικού και θεσμικού και στα πλαίσια της προσπάθειας να ενθαρρύνουμε όλους αυτούς τους αγωνιστές δημοκρατίας που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Γι' αυτό πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Για την ελευθερία και τη δημοκρατία ευχαριστώ πολύ. Σε όλους. May I just a, word? briefly.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 το, ο, τί κάνω, ναι, ναι, Vamos Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, που είναι η συζήτηση για την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ένωσης για το θέμα αυτό. Ο κύριος Παντζέρη για την πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης και μετά θα το συζητήσουμε. Κύριε Παντζέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι είναι αρκετά σαφή τα όσα προτείνονται ή τουλάχιστον ελπίζω ότι είναι. Ο στόχος που θέσαμε γράφοντας και αποστέλλοντας αυτά δεν είναι για να αντισταθμίσουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλαμε απλά και μόνο να διατυπώσουμε ορισμένες προτάσεις σε μια προσπάθεια να περάσουμε από μια περιγραφική λογική σε μια άλλη λογική. Προσπάθειά μας ήταν να υπάρξει μια αντιπαράθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τον ΙΠΑ, το εκπρόσωπο και τον ειδικό πεσταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και κυρίως ε, να ελέγξουμε και τη δική μας επιθυμία και την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη ορισμένων στόχων. Τα σημεία επί των οποίων επικεντρώθηκε η έκθεση αφορούν πρωτίστως, δεν θα αναφερθώ σε όλα λόγω έλλειψης χρόνου και εγώ θα προτιμούσα να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων. Το πρώτο σημαντικό σημείο και αντικείμενο της αντιπαράθεσης αφορά την ολοκλήρωση του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αναφορά στο άρθρο 21 το γεγονό ότι απαιτείται να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλε τι εξωτερικέ μα σχέσει χωρί να υπάρχει καμία εντελώ εξαίρεση. Θα πρέπει δηλαδή να γίνουν σημαντικά βήματα προ αυτή την κατεύθυνση. Για μα είναι σημαντικό κατ' ουσία να υπάρξει μια ημερησία διάταξη που θα αφορά αυτούς τους στόχους και όπου θα καταβληθούν προσπάθειες βεβαίως για την επίτευξή τους. Το άλλο σημαντικό σημείο που κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπογραμμιστεί αφορά την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην κοινότητα. Εκεί θα πρέπει να γίνει ένα ποιοτικό άλμα, γιατί περιορίζονται και στον, είπα το ειδικό πρόσωπο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα προσυπουγράψουν και οι άλλοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπή ε, και αυτό θα αφορά την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε άλλους τομείς, ας πούμε ε, θέματα μετανάστευση, εργασία, περιβάλλοντος, ε, διαχείρισης διαδικτύου, εμπόριο, επενδύσεις, τεχνολογία, επιχειρήσεις κτλ. Μία σειρά δηλαδή, σε μία σειρά από σημαντικού τομείς που θα πρέπει να υπάρχει πανταχικού παρουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να ανανεωθεί η εντολή του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητάμε να υπάρχει μια θεσμοθέτηση του ρόλου αυτού, της θέσης αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό για μας το να υπάρξει στη διάταξη του στρατηγικού πλάνου, του στρατηγικού σχεδίου, μια πλήρης εμπλοκή όλων των θεσμικών φορέων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών έτσι ώστε να, μπορέσει, ε, να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα ε, πράγματα στο μέλλον. Η έκθεση επικεντρώνεται σε μία σειρά από σημαντικούς τομείς. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στο γεγονός ε, ότι επικεντρωνόμαστε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή που αφορά και τις εμπορικές ε, σχέσεις που είναι υποδιαπραγμάτευση και εδώ είναι σημαντικό να αποκτήσουν κεντρικό ρόλο τα ανθρώπινα δικαιώματα και μην, αφορούν μόνο το θέμα των ελεύθερων συναλλαγών. Επικεντρωνόμαστε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφθοράς που είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Τονίζουμε το αίτημα του Κοινοβουλίου να υπάρξει δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διαφθοράς, την ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων ε, μηχανισμών, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαμε να δράσουμε. Θέτουμε το θέμα της ελευθερίας της ε, θρησκείας, της θρησκευτική έκφρασης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αναφέρομαι κυρίως ε, στη Μέση Ανατολή και στα όσα συμβαίνουν στη Συρία και το Ιράκ. Παράλληλα, θα ήθελα να αναφερθούμε στο θέμα δικαιωμάτων. Υπάρχει το σημαντικό θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Το θέμα αυτό το συζητήσαμε εκτενώς Όπως και το θέμα της απονομής του βραβείου Σάκαρον στον καθηγητή Νοβέ, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τους μαζικούς βιασμούς και τον βιασμό ως σημαντικό στοιχείο των ένοπλων συγκρούσεων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα της βίας που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά και ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός και εντός. Το θέμα των ε, λεσβιών, ε, των τρανσέξουαλ, ε, το θέμα των παιδιών, θέλουμε να υπάρχουν κοινά πρότυπα για την υποδοχή τους, την πληροφορίες που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Δικαιώματα των ατόμων με δικές ανάγκες, θέμα τεχνολογιών και διαδικτύου, ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο που αφορά τη δικαιοσύνη, τη διεθνή ε, δικαιοσύνη και ε, τα ποινικά θέματα, και θέματα σημαντικά που αφορούν τον ε, ε, τα βασανιστήρια και τις, ε, την καταδίκη σε θάνατο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω οικονομικοί πόροι, κυρίως για την προάσπιση αυτών που με τη σειρά τους προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό συμβαίνει παντού. Τέλος, η έκθεση θέλει να επικεντρωθεί κυρίως σε μια συγκεκριμένη θεματολογία, όχι σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και να μην χρησιμοποιήσει ένα περιγραφικό τρόπο, αυτό σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέματα επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και που πάντοτε αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε εκεί και να αφήσουμε κατά μέρο άλλα θέματα που αφορούν κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα το ρόλο των εξωτερικών αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου στις οποίες ε, ζητάμε να επιτελέσουν ένα ποιοτικό Άλμα, μιλώντας για τις ε, επισκέψεις που θα κάνουν στις διάφορες χώρες και τους ζητάμε να βάλουν στο κέντρο της προσοχής τους το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην ε, ε, ουσία θα πρέπει να εστιαστούν στα focal points των εξωτερικών αντιπροσωπιών. Με βάση λοιπόν αυτό θα έλεγα ότι βρίσκομαι εδώ για να ακούσω τους σκιώδεις εισηγητές, να ακούσω τι θα ήθελαν να πούν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι κατά κάποιο τρόπο να καταβάλει μια προσπάθεια να χαράξει μια πορεία που θα δώσει συνοχή στα όσα κάνουμε και θα μας δώσει τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε κατά πόσον οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι επιτεύξιμοι. Εδώ δεν θα πρέπει απλά και μόνο να αναλωθούμε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα πρέπει να επιτελέσουμε ένα ποιοτικό άλμα. Αυτό αφορά εμάς και αφορά και τον είπα το εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκα συντάσσοντας αυτή την έκθεση. Είμαι στη διάθεσή σας τώρα για να ακούσω τι έχετε να μου πείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Να δώσω το λόγο στους Κιώδης Πρώτος ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον συνάδελφο κύριο Παντσέρη για το εξαιρετικό σχέδιο εκθέσεως που μόλις μας παρουσίασε. Εκτίμησα όλος ιδιαίτερος τη συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που οργάνωσε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών αυτών οργανώσεων ε, που παρέστησαν και έκαναν πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Όσον αφορά τώρα το κείμενο του συγκεκριμένου ψηφίσματος, Έχω κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες μπορεί να μετατραπούν σε τροπολογίες. 15 τροπολογίες υποσχέθηκα στον κύριο Παντσέρη και ελπίζω να μπορέσω να τηρήσω την υπόσχεσή μου. Πέρα όμως από τα αστεία, ελπίζω να έχουμε ένα καλό κείμενο το οποίο θα τύχει υπερψήφισης ε, και στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια. Τα σχόλιά μου τώρα. Να αρχίσω με μία παρατήρηση σε σχέση του τι συμπεριλαμβάνει ο τίτλος «Ευρωπαϊκή πολιτική για την υποστήριξη του εκδημοκρατισμού και των δημοκρατικών εκλογών». Δύο παρατηρήσεις για να ενισχύσουμε αυτή την ιδέα του εκδημοκρατισμού. Φυσικά οι εκλογικές πτυχές είναι πάρα πολύ σημαντικές, τονίζονται παρκώ στο κείμενο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνουν με περισσότερες αναφορές. Δηλαδή, συγκεκριμένα τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να προχωρήσει μια δημοκρατική κοινωνία και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει μια τέτοια διαδικασία. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία συνοχής ως προς τις δικές μας δράσεις και μιλάω για τις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Ζητούμε συνοχή από όλους τους υπόλοιπους εταίρους, αλλά πρέπει να επιμείνουμε και εμείς οι ίδιοι να είμαστε συνεκτικοί. Οι δραστηριότητες της Επιτροπής, Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν πρέπει να, να επικαλύπτονται με τις ε, δραστηριότητες Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ επίσης συντάσσει μια ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θέματα όπως το δημοψήφισμα στην Κροατία, η νομοθεσία, πρόσφατη νομοθεσία στην Λιθουανία ή ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στη δική μας έκθεση. Πιστεύουμε ότι, πιστεύω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία οι συνάδελφοι της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ε, πρέπει να αναλάβουν. Νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν ε, στο πλαίσιο της δικής τους επιτροπή. Δεν θα πρέπει να επιμένουμε εμείς σε αυτό. Δεν θα πρέπει δηλαδή να χάνουμε εμείς ε, τη δική μας εστίαση ε, εξετάζοντας θέματα που ανήκουν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Τώρα, σε σχέση με το σχέδιο ψηφίσματος του κυρίου Παντσέρη, στην παράγραφο 9 θα ήθελε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΙΕΔ μία έκθεση εφαρμογή σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για το 2013. Νομίζω ότι η ετήσια έκθεση για τη δημοκρατία ούτως ή άλλως επιτυγχάνει αυτό το σκοπό. Θέλουμε να ζητήσουμε να επανεπισημανθεί δηλαδή κάτι το οποίο έχει ήδη αναφερθεί στην έκθεση. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε την έκθεση αυτή, την ευκαιρία να συζητήσουμε την έκθεση αυτή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ζητήσουμε μία ακόμη έκθεση, μία έκθεση εφαρμογής όπως προτείνει η παράγραφος αυτή η παριθμόν 9. Όσον αφορά τώρα τις διοργανικές σχέσεις, να επιμείνω σε κάτι και θα ήθελα να εισαχθεί μια νέα παράγραφος, ότι δεν έχουμε λάβει γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ψήφισμα που μόλις εγκρίναμε για το 2012. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Μια γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να λάβουμε. Είναι ένα είδος συνεργασίας διοργανικής και μάλιστα πολύ σημαντική μορφή συνεργασίας και πιστεύω ότι η γραπτή απάντηση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από συζήτηση στην Ολομέλεια. Η συζήτηση στην Ολομέλεια είναι βεβαίως απαραίτητη, αλλά είναι πολιτική συζήτηση, ενώ μια γραπτή απάντηση δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, επιληφθεί όλων των θεμάτων που έχουν αναφερθεί στην ετήσια έκθεση. Συγκεκριμένα για την αντίθεση έκθεση για το 2012 μιλάω. Και θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου, γιατί δεν μας έχει στείλει γραπτή απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάπως περίεργο είναι ότι δεν μας έχει στείλει γραπτή απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως δεν έλαβε το αίτημά μας. Ένα ακόμη σχόλιο σε σχέση με την παράγραφο 14 αυτή τη φορά. Η παράγραφος 14 προτείνει να έχουμε κοινά πρότυπα για τα κράτη-μέλη και τους αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν γίνονται αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους στρατηγικούς εταίρους της. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες και πρέπει να αναλύσουμε και τα προφίλ των ε, εταίρων μας για να είμαστε αποτελεσματικοί. Παράγραφος 28. Εκεί μπορούμε νομίζω να εκφράσουμε το ότι μας ε, λυπεί το γεγονός ότι μέχρι το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε αντιπροσωπεία που να το εκπροσωπεί ε, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στη συγκεκριμένη παράγραφο ότι μιλάμε για τη συνεργασία με αυτό με αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό οργανισμό και πρέπει να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας πάρα πολύ ε, σαφώς. Όσον αφορά τώρα το τμήμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, πολιτική βοήθειας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αρκεστούμε σε μία παράγραφο και σε ένα πρόβλημα λέει ότι καλούμε ε, για συντονισμένη ε, ε, διαχείριση του προβλήματος της αρπαγής γης. Μόνο γι' αυτό μιλάμε εδώ, αυτό το πρόβλημα, σε αυτό το πρόβλημα αναφερόμαστε. Ο μόν, ως μόνιμος εισηγητής για τις αναπτυξιακές πολιτικές, με ανησυχεί αυτό το θέμα. Ίσως θα έπρεπε να εισαχθούν και άλλες παραγράφ, παράγραφοι για να μπορέσουμε να καλύψουμε το ευρύτερο θέμα της αναπτυξιακής ενίσχυσης. Όσον αφορά τώρα το συντονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δύο σχόλια έχω. Πρώτον, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών ε, των αντιπροσωπιών. Νομίζω ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν ήδη και είναι καλές. Νομίζουμε όμως ότι χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή και ενισχυμένη συνεργασία σε εσωτερικό επίπεδο. Προσωπικά πιστεύω ότι μια περιεκτική γραπτή έκθεση δεν θα μας βοηθήσει. Χρειαζόμαστε μια καλή πολιτική συνεργασία στο, στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι αυτό είναι δυνατό. Όσον αφορά τώρα κατεπήγοντα ψηφίσματα, έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Χρειαζόμαστε μια διαδικασία που να μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί στην Ολομέλεια το ψήφισμα και έχουμε ήδη κάνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Ίσως θα μπορούμε να αναφερθούμε και στην έγκριση ενός παραρτήματος στην έκθεση που θα ε, συμπεριλαμβάνει τον, ε, ε, τους πολιτικούς εχμαλώτους σε όλο τον κόσμο ένα διεξοδικό κατάλογο και για να μην γίνουν σφάλματα, ίσως θα έπρεπε ο κατάλογος να συμπεριλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που έχουμε εμεί συζητήσει στα δικά μας κατεπήγοντα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλύτερη λύση από το να έχουμε ένα διεξοδικό κατάλογο με πολιτικούς εχμαλώτους, πολιτικούς κρατουμένους. Νομίζω ότι το παράδειγμα αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μία λύση. Όλες οι περιπτώσεις που έχουν ε, επισημάνει οι δικές μας πολιτικές ομάδες ε, μέσω ε, ψηφισμάτων στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι μπορούμε να διχειριστούμε καλύτερα ένα τέτοιο κατάλογο και έτσι θα είχαμε πολύ καλύτερη συμπεριφορά κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα παίρνουμε δηλαδή απλώς ονόματα από τους καταλόγους άλλων ανθρώπων, θα ε, έχουμε τα δικά μας ονόματα τα οποία θα αναφέρουμε. Υποθέτω ότι και άλλοι συνάδελφοι θα έχουν ε, συστάσεις και επίσης θα ε, υποβάλλουν τροπολογίες προκειμένου να καλυφθούν θέματα όπως η ελευθερία της θρησκείας, της έκφρασης. Θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο για το πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε καλύτερα τη θέση ε, του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριος Χέγκελ. Είμαι νέος ευρωβουλευτής. Αλλά δεν ε, άρχισα τώρα να ασχολούμαι με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είμαι μέλο τη διεθνού Αμνηστία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια από πλευρά τη ομάδα μα για την έκθεση αυτή. Πρώτον, συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή ότι η έκθεση αυτή σε μεγάλο βαθμό επαναλαμβάνει αυτά που λέγονται και σε άλλες επιτροπές. Ανέφερε τη ΛΥΜΠΕ για το θέμα της Κροατίας. Συμφωνώ πλήρως με τη θέση του. Αλλά έχω μια γενικότερη αντίρρηση για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι διευρύνουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε θέματα που δεν σχετίζονται καθόλου με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ελάχιστα. Παράδειγμα. Δεν το πίστεψα όταν το είδα. Υπάρχει η σύσταση ότι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρέπει να εισαχθεί στην Ευρώπη. Ε, μα τι σημαίνει αυτό. Τι σχέση έχει την ανθρώπινα δικαιώματα. Αν πραγματικά εγκριθεί αυτή η παράγραφος, τότε γιατί να μην πούμε ότι πρέπει να καταγγείλουμε και την υπερβολική φορολογία. Και αυτό είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα δεν είναι δυνατόν τώρα τέτοιες ε, πολύ στενά πολιτικές απόψεις ε, να βαφτίζονται ανθρώπινα δικαιώματα και να περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια προσέγγισης σε αυτή την έκθεση. Και τι σημαίνει αυτό για όλους αυτούς που υποφέρουν από βασανιστήρια, ε, που είναι στη φυλακή αδίκως, που απειλούνται ε, με δολοφονία. Εάν προβάλλουμε τέτοιες ε, στενά πολιτικές ιδέες που δεν έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Σας παρακαλώ λοιπόν, κάνω έκκληση να εστιάσουμε στα θέματα που είναι πραγματικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να μην επιτρέπουμε την πολιτική μας προσέγγιση να επισέρχεται. Επίση, η έκθεση αυτή δεν σέβεται την επικουρικότητα. Θα θυμάστε όλα αυτά που είπε ο Γιούνκερ και οι περί αυτών. Μας λένε ότι η επικουρικότητα πρέπει να είναι πάντα στο μυαλό μας. Ακόμη και ο Πάπας τόνισε πόσο αναγκαία είναι η επικουρικότητα. Δυο φορές το είπε. Αλλά αν διαβάσετε την έκθεση θα δείτε να αναφέρει πολλά που δεν είναι θέμα ενωσιακής αλλά εθνικής αρμοδιότητας. Επίσης ε, προωθούνται και θέματα οικογενειακής πολιτικής. Υποτίθεται ότι είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε αυτό σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά, οι διακρίσεις ε, σε βάρος των ατόμων ε, LGBTI πρέπει να αναφερθούν. Αλλά αυτή η αντίληψη ότι όλες οι χώρες πρέπει να εφαρμόσουν ε, το γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται. Αυτό είναι θέμα εθνικού δικαίου. Βεβαίως, καταπάτηση των δικαιωμάτων των μεταναστών να συμπεριληφθεί. Αλλά δεν θα πρέπει να συζητήσουμε συνολικά το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Η διαφθορά είναι τρομερό πρόβλημα. Μα, αλλά γιατί πρέπει να αναφερθεί σε μια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ως ομάδα, εμείς ως ομάδα επίσης διαφωνούμε για το θέμα της θανατικής ποινής. Εγώ διαφωνώ με ορισμένα μέλη της ομάδας μου ότι σε μια δημοκρατική χώρα δεν πρέπει να επικρίνουμε τη θανατική ποινή. Εφόσον επικρίνουμε και καταδικάζουμε τα βασανιστήρια, πρέπει να καταδικάζουμε και τη θανατική ποινή για όλα τα καθεστώτα, δημοκρατικά ή όχι. Οπότε θα υποβάλουμε μια σειρά από τροπολογίες και σας καλώ και αυτό είναι το κύριο που θέλω να πω. Να επανέλθουμε και πάλι στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τους ανθρώπους των οποίων παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην χρησιμοποιούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για να περάσουμε την πολιτική μα άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάνκελ. Ο κύριος Οστσεβίτσιους. Ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεση του συναδέλφου μας Κύριο Παντσέρη στοιχίζεται πολύ καλά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό μας βοηθάει. Μας βοηθάει να έχουμε μια έκθεση συνοπτική που να δίνει ένα σαφές μήνυμα. Και μας επιτρέπει να μην ασχοληθούμε με τις 150 εθνικές στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναφέρει η έκθεση του Συμβουλίου. Τώρα κάποια σχόλια και προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν το κείμενο. Έχουμε βέβαια κάποιες ε, προόδους και κάποιες ε, επιδεινώσεις και κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ε, που θα πρέπει να αναφερθούν λοιπόν για κάποιες χώρες. Να αναφέρουμε και τα επιτεύγματα, της προόδους κάποιων χωρών. Αυτό θα ενεθάρρυναν τις χώρες αυτές να συνεχίσουν την θετική τους πορεία. Δεν θα πρέπει να αναφέρουμε πολλές βέβαια, αλλά να επιλέξουμε τα καλύτερα παραδείγματα όπου θέλουμε να δείξουμε ότι εκτιμούμε αυτά που επετεύχθησαν για να τα προωθήσουμε περαιτέρω. Έχουμε εδώ την παράγραφο για τη θανατική ποινή. Γιατί να μην αναφερθούμε στις πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις λοιπόν και για θανατική ποινή όπου έχει υπάρξει πρόοδος και για άλλα θέματα. Ο διάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ετήσια έκθεση αναφέρει ότι είχαμε για πρώτη φορά τέτοιο διάλογο με τη Νότια Αφρική και τη Βόρεια Κορέα. Γιατί να μην το ξαναπούμε. Το είπαμε πρώτη φορά στην ετήσια έκθεση για το 2013. Έτσι θα γίνει πιο συγκεκριμένη η έκθεση και όχι απλώς παραθετική. Δεύτερον, λείπουν ορισμένα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση του Συμβουλίου. Αλλά όχι εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι περιορισμένο το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες αναφορές σε μειονότητες και εγχώριους πληθυσμούς, ηθαγενείς πληθυσμούς. Θα έπρεπε να αναφέρονται. Τουλάχιστον οι ηθαγενείς πληθυσμοί θα πρέπει να αναφερθούν σε σχέση με την αρπαγή γεών και οι μειονότητες. Γιατί μιλάμε μόνο για τις θρησκευτικέ μειονότητες. Υπάρχουν εθνικές, πολιτιστικές μειονότητες. Τέλος, τέλος. Για να διαφοροποιήσουμε την έκθεση του Συμβουλίου από την, συγγνώμη, του Κοινοβουλίου από την έκθεση του Συμβουλίου, να μην είναι απλώς μια συνόψηση της έκθεσης του Συμβουλίου, πρέπει να αναφερθούμε στη δραστηριότητα του Κοινοβουλίου. Το τελευταίο, τελευταίο τμήμα της έκθεσης αναφέρεται στην ε, δουλειά που κάνει το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι λίγο πιο εκτεταμένη και να περιλάβει και άλλα θέματα. Να σημειώσει αυτά που έχουμε κάνει μέσω των κατεπηγόντων για να βελτιώσουμε την προστασία των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, είχαμε πρόσφατα μία κρόαση για τον Μπαχρέιν και χρειάζεται πιο έντονη δημόσια διπλωματία. να κάνουμε κάτι σαν αυτό που έκανε ο εισηγητής κύριος Ντόνσκης το 2011 να επισυνάψουμε ένα παράρτημα για την δραστηριότητα του Κοινοβουλίου μας. Αυτό θα εμπλούτιζε την έκθεση ουσιοδός. Τέλος και καταληκτικά και συμπερασματικά. Νομίζω ότι είναι καλό σημείο κίνησης αυτό το σχέδιο έκθεσης. Θα υποβάλουμε τα σχόλια και τις τροπολογίες μας εν ευθέτω χρόνο. Σας υπόσχομαι ότι θα είναι λιγότερες από 50. Προσβλέπω στην επόμενη συνεδρίασή μας να έχουμε μία συζήτηση συντονισμού για να καταλήξουμε σε μία θαυμάσια έκθεση που νομίζω ότι μπορούμε να ε, συντάξουμε. Ο κύριος Ροκμπίλερ, η κυρία Ροκμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έριξα ένα ματιά στην έκθεση του κυρίου Κούκαν. Υποβλήθηκαν 76 τροπολογίες. Σας υποσχέθηκα, κύριε Παντσέρη, ότι δεν θα τις ξεπεράσουμε. Θα ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό, αλλά δεν φανταζόμουν πόσες θα, θα υπέβαλα εγώ. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή έκθεση. Κάνετε μία αναφορά στους πρόσφυγες, ε, αναφέρεστε στο κόστος της μη συμμόρφωσης με τα όσα προβλέπονται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν επίσης συστάσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να κάνει το Κοινοβούλιο. Και ο κύριος Σοστρεβίτσι και ο κύριος Πρέντα αναφέρθηκαν στα σημεία αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία πιο εκτενή παράγραφος. Και θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο στρατηγικό έγγραφο σχετικά με το τι κάνει ακριβώς, το, τι κάνουν τα κοινοβούλια. Γίνεται ή θα πρέπει να γίνει. Ετήσια έκθεση. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε. Η ετήσια έκθεση είναι μια έκθεση 800 σελίδων και βεβαίως θα φανταστείτε ότι δεν την έχω διαβάσει. Ε, ε, το ερώτημά μου στους συναδέλφους και στη γραμματεία, το διαβάζετε τη διαβάζετε. Αυτή την έκθεση διαβάζετε απλά και μόνο στις παραγράφους που σας ενδιαφέρουν. Υπάρχει μια ευρύτερη ιδέα εδώ. Έχει άμεση σχέση για την πολιτική που εφαρμόζουμε εμείς, βεβαίως μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς. Αλλά ενδεχομένως στο μέλλον θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάθε χρόνο να συντάσσεται μια στρατηγική ευσύνοπη έκθεση σχετικά με το τι έχει εφαρμοστεί, τι έχει επιτευχθεί, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, στην περίπτωση αυτή είναι μάλλον παράλογο. Ήταν χρονιά εκλογών. Ζητάμε μια έκθεση την οποία ε, γράφεται το, συντάσσεται το 2013 και την υιοθετήσουμε το 2014. Και περιοριζόμαστε και δεν μιλάμε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, αν έχει κάποιο νόημα να υποβάλλεται μια τόσο εκτενή έκθεση. Είπατε, αναφέρατε το σημείο 6 της ετήσιας έκθεσης ή μάλλον εκφράζεται το αίτημα να εξεταστούν οι εκθέσεις ε, των χωρών. Δεν ήταν σαφές αυτό. Στην παράγραφο 9 έχουμε τις στρατηγικές των χωρών. Χρησιμοποιούνται όλοι αυτοί οι δείκτες και μπαίνουν υπό το 6. Αυτές οι εκτέσεις ε, είναι πολύ μικρές. Ε, δηλαδή ζητάμε από το ιερές να ε, διπλασιάσει τις προσπάθειες του κάπου κάνει και να αποφευθεί αυτό. Εμείς εστιαζόμαστε στη στρατηγική των χωρών, εκεί που υπάρχουν αυτοί οι δείκτες και εμείς ζητάμε πρόσβαση σε αυτούς. να εξετάσω μερικές από τις τροπολογίες. Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την 53, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να λέμε ότι η πλειοψηφία των κονδυλίων δίνονται στους ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ποσοτικά αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι χαιρετίζουμε τον νέο κανονισμό, αλλά μας δυσαρεστεί το γεγονός ότι γίνονται περικοπές των κονδυλίων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ένα περισσότερο ελαστικό τρόπο. Ένα ερώτημα για τον είπα το εκπρόσωπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον ειδικό εισηγητή. Στο σημείο 13 αναφέρατε, λέτε ότι υπάρχει ένα αίτημα θεσμοθέτηση της θέσης ε, του ειδικού απεσταλμένου έτσι ώστε να, να είναι μόνιμη αυτή η θέση. Ερώτηση. Δεν θα πετύσει αυτό αλλαγή στις συνθήκες. Όντως πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι μόνιμη αυτή η θέση. Παράγραφος 79 στα καταπήγοντα και βραβείο Σαχάροφ. Πώς θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει και ένα θέμα που αφορά την ε, Frontex και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ύστερα την ανάγκη για την ε, δημιουργία ενός πλαισίου που αφορά το εμπόριο ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μας στην Τρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ζητήσει και η κυρία Χιμένεθ Μπεθερίλ το λόγο. Είστε από πλευράς της Επιτροπής Ανάπτυξης, ε, η συντάκτης ε, της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Να συγχαρώ τον κύριο Παντσέρη για την έκθεσή του που είναι τόσο πλήρης. Προσπαθεί να συνοψίσει και να καθορίσει προτεραιότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μια ολόκληρη χρονιά οι παρεμβιάσεις είναι τόσο πολυάρθμες και σε τόσο πολλές χώρες που θέλει πολλή δουλειά για να τα συμπεριλάβει κανείς όλα σε μια έκθεση. Πρέπει όμως να στοχάσουμε σε αυτό που θεωρούμε παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συμφωνώ λοιπόν με κάποιους συντρόφους που είπαν ότι ορισμένα είναι θέματα λίμπε. Είμαι και στη λίμπε. Γιατί είναι θέματα που αφορούν την ένωσή μας. Συμφωνώ με τη σημασία που αποδίδει ο εισηγητής στην εξωτερική μας πολιτική οι οικονομικές μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές, όπως ακούσαμε και στην προηγούμενη ακρόαση. Αλλά βέβαια οι οικονομικές σχέσεις δεν θα υπήρχαν εάν δεν υπήρχαν άτομα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οπότε η αξιοπρέπεια αυτή πρέπει να υπερέχει των οικονομικών σχέσεων. Πολλές φορές κατά τις συζητήσεις με τις αντίστοιχες ε, αντιπροσωπείες ε, κάποιων χωρών ή όταν συζητάμε για συμφωνίες και αναθεώρηση συμφωνιών βλέπουμε ότι υπάρχουν μια πολύ στενή αντιμετώπιση. Διότι το πιο σημαντικό για κάθε χώρα που έχει προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της χώρας αυτής, αλλά παράλληλα να προωθήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίω, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για του αγωνιστέ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Και επίση συμφωνώ με τον κεντρικό ρόλο που αποδίδει στα δικαιώματα των γυναικών, που είναι το πιο ευάλωτο τμήμα τη κοινωνία. Σε πολλέ χώρε βλέπουμε. Βλέπουμε ότι για παράδειγμα ο βιασμός χρησιμοποιείται ως όπλο στον πόλεμο, επίσης ε, η εμπορία ανθρώπων που σχετίζεται και με τη μετανάστευση, η σεξουαλική εκμετάλλευση που έχει να κάνει και με τις γυναίκες και με τα παιδιά και βεβαίως και για τα θέματα των παιδιών, για τις, τους υποχρεωτικούς γάμους, για τις, τους γενετικούς ακροτηριασμούς. Συμφωνώ με όλα αυτά. Και επειδή είμαι από την Επιτροπή Ανάπτυξης, θεωρώ ότι πρέπει να εμβαθύνουμε για ορισμένα θέματα. Θα συνεργαστούμε γι' αυτό. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που το αναφέρετε, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να επεκταθείτε, είναι η ασφάλεια και η σωστή διακυβέρνηση. Είναι η βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να μιλήσουμε για τις καταστάσεις πολέμων και για την τρομοκρατία που βλέπουμε πόσες χιλιάδες θύματα προκαλεί. Πρέπει να αναφερθεί πιο εκτεταμένα και θα το αναφέρω στις τροπολογίες που θα υποβάλω. Μιλήσατε για την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα, θέματα, για τα θύματα ε, βιασμών και βίας. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη πρέπει να αφορά όλα τα θύματα όχι μόνο τα θύματα που αναφέρατε. Είναι κάτι πολύ γενικότερο. Αυτά σας συγχαίρω για την έκθεση αυτή, ε, την οποία θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε όπου θεωρούμε σκόπιμο. Ευχαριστώ. Η κυρία Τάισεν, Ελίζαπεθ Τάισεν, που είναι επικεφαλής ε, του Τμήματος για Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, για ε, την έκθεση του κυρίου Παντσέρη. Ε, ακούσαμε πολύ προσεκτικά αυτά που είπε Ήρθαμε σε επαφή με το προσωπικό σας και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνούμε με τη θεματική προσέγγιση, όπως επίσης και με την επιλογή και τη δομή ε, των θεμάτων. Επίσης, συμφωνούμε με τη γενική αρχή στην οποία αναφέρεστε την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια στην εφαρμογή των πολιτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επίσης και την ενίσχυση εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής. Αυτή η αρχή, από κοινού με την η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων, είναι η βάση του στρατηγικού μας πλαισίου, που θα αποτελέσει ευρύτερη αρχή για μας που θα μας καθοδηγήσει και το νέο ε, πρόγραμμα δράσης. Για το νέο αυτό πρόγραμμα ε, περιμένουμε την έγκριση της κυρίας Μουγκερίνη, αλλά έχουμε αρχίσει την προπαρασκευαστική μας εργασία, από την, ε, όπως το γνωρίζετε από την προηγούμενη μας συζήτηση, οπότε υποστηρίζουμε τις προσπάθησε σας και ελπίζουμε να επικεντρωθείτε στην ιεράρχηση των δραστηριοτήτων αλλά να μην μειώσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας ειδικότερα όσον αφορά την ενσωμάτωση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε πολιτική. Επίσης να επιβεβαιώσω ότι έχουμε αρχίσει την προπαρασκευή της ετήσιας έκθεσης του 2014. Θα ακολουθήσει την ίδια μορφή με τα προηγούμενα έτη, ένα θεματικό τμήμα που αφορά τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης και μετά ένα γεωγραφικό τμήμα που καλύπτει όλες τις περιφέρειες και όλες τις χώρες. Η, το 2000, η εκθέση του 2014 θα δώσει μια ανάλυση των προτεραιοτήτων μας και η αξιολόγηση αυτών θα μας καθοδηγήσει στην, ε, στον προγραμματισμό του νέου ε, προγράμματος δράσας, δράσης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθάτε στις προσπάθειές μας ε, και θα επανέλθω για το, για το θέμα αυτό όταν θα έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο εκθεσής σας. Επίσης για τις θεματικές πολιτικές θα έπρεπε ίσως να τονίσουμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την εφαρμογή των μέσων που έχουμε επιτόπου. Οι συστάσεις σας ε, συμφωνούν με την ε, δική μας συλλογιστική, δηλαδή και εμείς πιστεύουμε ότι οι κατευθυντήρες γραμμές πρέπει να ε, μεταγράφονται καλύτερα σε συγκεκριμένες δράσεις και για να γίνει είμαστε πεπισμένοι όπως και εσείς ότι πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση όπως επίσης και την ενίσχυση της θέσης των σημείων ε, εστίασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα διάφορα κράτη-μέλη, ώστε να ε, μπορούν να ε, αξιοποιούν καλύτερα την, τις καλύτερες εμπειρίες και πρακτικές. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την διαδικασία έγκρισης της έκθεσης αλλά και των τροπολογιών. Θα ήθελα να κάνω σχόλια για τρεις, παρατηρι... για παραγράφους. Πρώτον, παράγραφος 6 και παράγραφος 9. Επικροτούμε τα σχόλια της κυρίας Λοχ Μπίλερ για τις προτεραιότητες και τους δείκτες. Συμφωνούμε, ε, όπως είπα, θα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση για το νέο ε, σχέδιο δράσης, χωρίς να ξεχάσουμε εξετάσουμε ε, την προσέγγισή μας ε, για όλες τις θεματικές ενότητες. Όσον αφορά όμως ε, τους πίνακες αξιολόγησης και τους δείκτες, σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να είναι οι επιδόσεις μας μετρήσιμες και όπως γνωρίζετε έχουμε γκρίνει ένα πρόσφατο έγγραφο που θα μπορούσε να καθοδηγήσει την ε, προσέγγισή μας σε διάφορους τομείς. Θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε την ευκαιρία στον εκπρόσωπό μας να αξιολογήσει ε, ε, τον πίνακα αξιολόγησης και τους δείκτες και θα επανέλθουμε από αυτού. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στο σημείο ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρήσεις. Θα ήθελα να πω, ίσως να το γνωρίζετε, ότι το θέμα αυτό ότι υπάρχει ένα φόρουμ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή στη Γενέβη ε, το οποίο, στο, στο, στο οποίο συμμετέχει και δικό μας προσωπικό από την ΕΕΔ. Ξέρετε ότι είχαμε μια συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις στη Γενέβη και υπήρχαν και δύο ψηφίσματα για το θέμα αυτό. Επικροτούμε το γεγονός ότι ο απότερος στόχος είναι να έχουμε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο, αλλά για την ώρα ενισχύουμε και υποστηρίζουμε πλήρως ε, το, το, την αρχή ε, καθοδήγησης του ΟΗΕ, το οποίο, η οποία εγκρίθηκε μετά από πολύ μακροχρόνιες διαδικασίες, ε, μετά από ε, προάσπιση ε, των, ε, μετά από μεγάλες προσπάθειες προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ. Ίσως πρέπει λοιπόν το δεύτερο τμήμα της παραγράφου, όταν μιλάτε για τα νομικά δεσμευτικά μέσα, να το χρωματίσετε λιγάκι, γιατί όταν μιλάμε για τη σχέση μας με την Νότια Αφρική, για παράδειγμα, έχουμε διμερείς, έχουμε διμερείς επαφές με τους εταίρους μας, Προσπαθούμε λοιπόν να προσαρμόσουμε την προσέγγιση μας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξακολουθούμε να είμαστε άνοιχτοι και ε, αν χρειαστεί θα ε, κάνουμε μερικά ακόμη σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο πριν ε, επανέλθει ο κύριος Παντσέρη. Όχι. Ο κύριο Σέντε δυστυχώ απουσιάζει και θα ήθελα να του παραπέμψω και πάλι την ιδέα της ιδεολογικής προσέγγισης. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι πολιτικό. Ενδεχομένω θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα τι ακριβώ εννοούμε τον όρο ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν από μερικά χρόνια, ο αρχιτέκτονας Βέι Βέι αν θυμάστε, ήταν γνωστό γιατί σχεδίασε την ε, Φωλιά του πουλιού στο ε, στάδιο του Πεκίνου. Μετά από την αποφυλάκησή του είπε ότι θα μετανιώσετε για τη σιωπή σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν όλα αυτά πνιγούν μέσα στα τα χρήματα, θα ε, μετανιώσετε κάποια στιγμή. Και βλέπετε ότι κάνει μια άμεση αναφορά στο θέμα της, ε, των χρημάτων. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την προσέγγισή μας, θα ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε ποιος είναι ο μύτος που συνδέει τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως σχετικά με το Χονγκ Κόνγκ, με την νεαρή έφηβη στο Ιράν, με τις γυναίκες του ε, Ιράν που επιμένουν να οδηγούν ένα αυτοκίνητο. Τι ενώνει τον κάποιον που εργάζεται σε μια επιχείρηση και τον απειλούν με απόλυση τον παράνομο εργάτη τι σχέση υπάρχει μεταξύ την προσβολή της δημόσιας εικόνας της γυναίκας των αυταρχικών νόμων που αφορούν τις βιολογικές διαθήκες, τους κανονισμούς για την ομοφομιδία, τους κανόνες που δεν υπάρχουν και την αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ' ουσία πιστεύω ότι ο κοινό παράγοντας που ενώνει όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν την ε, ε, ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, το φύλλο κτλ. Κατ' ουσία αυτή είναι η δική μου άποψη. Η πραγματική πρόκληση στον κόσμο για μας είναι το να δεχτούμε την πρόκληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολό τους, πολιτικά, κοινωνικά, ανθρώπινα δικαιώματα ως βάση για μια νέα οικονομία που θα καταλήξει σε μια δημοκρατία πολιτισμού θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε χώρα. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση, δεν είναι ιδεολογική προσέγγιση. Θα έλεγα ότι είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις όλων των βουλευτών γιατί αν ο στόχος είναι να είμαστε πιο φιλόδοξοι, νομίζω ότι θα πρέπει να τον θέσουμε αυτό το στόχο προσπάθεια να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι. Τώρα για να φερθώ πρακτικά στα θέματα που εφήγησαν. Κρίστιαν Μπρέντα, πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία παράγραφος περισσότερο έντονη σε ό,τι αφορά τη στήριξη στη δημοκρατία και στο θέμα των εκλογών να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντρεώσει αυτές τις, αυτή τη δημοκρατική μετάφαση. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας το κατά πόσον θα πρέπει να ενδιαφερθούμε για όσα κάνει η Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων. Ερωτηματικό. Θέλω να το συζητήσουμε. Γιατί τη στιγμή κατά την οποία ζητάμε να υπάρχει συνοχή μεταξύ τη εξωτερική και τη εσωτερική δράση, θα πρέπει να γίνει κάποια μνήμα. Γιατί αν ζητάμε, απλά, αν λέμε απλά και μόνο να αποφύγουμε να υπάρχουν νόμοι που οδηγούν ε, του ομοφυλόφιλου στην Ουγγάντα στη φυλακή, ενώ στην Ευρώπη υιοθετούνται νόμοι που κατά το μάλλον ή τον θέτουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να θέσει ένα θέμα συνοχής ή μάλλον συνέπειας. Ε, ε, γιατί ε, θα έλεγα ότι είναι μια αντίφαση που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να, αντιμετωπίσουμε. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά το σημείο 14 και το σημείο 28 που αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη. Κανένα πρόβλημα να διευρύνουμε και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης. Γιατί είναι αλήθεια ότι επικαιρωνόμαστε μόνο στο θέμα της υφαρπαγής των γεών ένα θέμα που αφορά την υποεπιτροπή των δικαιωμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βασικές γραμμές με τις αντιπροσωπίες, θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα τη στιγμή κατά την οποία η υπηρεσία εξωτερικής δράσης εντόπισε τα εστιακά σημεία μέσα στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητο και για μας να είμαστε συνεπείς και να θέσουμε νέες γραμμές τις οποίες θα βασίσουμε τις μελλοντικέ μας εργασίες για αυτά τα focal points και από εκεί και η ανάγκη να τροποποιήσουμε λίγο τη στάση μας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το αντίθετο, το αντίθετο θα έλεγα ότι θα πρέπει να βρούμε τις πλέον κατάλληλες διατυπώσεις για να ενδυναμώσουμε το κεφάλαιο αυτό αναφερόμενοι σε όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως Κοινοβούλιο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξωτερική δράση. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του κυρίου Αντερβίσιους, ναι, ενδεχομένω θα πρέπει να πούμε κάτι για τις τοπικές μειονότητες. Ναι, θα παρέμβω και εγώ γιατί αυτό σε ό,τι αφορά τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα και τις κάστες και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Εξάλλου, το είπα όχι σήμερα, αλλά στην τελευταία συνάντηση, ότι θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε ορισμένα γεωγραφικά παραδείγματα που θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε, όχι όμως να επαναλάβουμε τη μία χώρα μετά την άλλη. Αυτό είναι ένα θέμα περιγραφικό, δεν είναι πλέον χρήσιμο. Συμφωνώ ε, να τονίσουμε περισσότερο ε, αυτό το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ απόλυτα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει και ένα στρατηγικό σχέδιο που θα, εγκριθεί, θα συζητηθεί και θα ε, εγκριθεί στην Ολομέλεια για να υπάρξει μια μεγαλύτερη δέσμευση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράγραφος 6-9 η παραπράγραφη 6-9, η διπλή εργασία. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ο στόχος που θα πρέπει να θέσουμε είναι ότι τη στιγμή κατά την οποία δημιουργούμε μια στρατηγική για κάθε χώρα, αυτή επί, επί, η Επιτροπή του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ελέγξει την πορεία των εργασιών. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να παραμένουν μόνο θέματα επιχάρτου. Υπάρχει και η δυνατότητα μιας κατηδίαν συζήτησης σχετικά με την πορεία των εργασιών. Το ζητούμενο είναι πώς είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι των διαφόρων στρατηγικών. Πιστεύω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ειλικρινά δεν ξέρω ε, αν θα πρέπει να ε, συζητήσουμε το θέμα του ε, μόνιμου εκπροσώπου σε σχέση με τις συνθήκες. Τι να πω, καλύτερα να μην τις αγγίζουμε τις συνθήκες. Εγώ δεν αμφισβητώ τη θεσμοθέτηση του ρόλου ενδεχομένως ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο λειτουργία. Ο στόχος που θα πρέπει να θέσουμε είναι ο ειδικό ε, εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για μας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε μέσα σε ένα χρόνο. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει μια διαρκή παρουσία και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το έχει μονίμως κατά νου. Πιστεύω ότι απάντησα, θα έλεγα, σε όλα τα ερωτήματα που ετέθεσαν. Όσο λιγότερες τροπολογίες, τόσο καλύτερα βέβαια. Για σας το λέω, για να μην κουράζεστε. Ύστερα ε, Εμπιστευτείτε με. Ας γράψουμε από κοινού μια έκθεση που θα είναι χρήσιμη και σε εμά και στους άλλους, δηλαδή στην κοινωνία των πολιτών που κατά κάποιο τρόπο συνέβαλαν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ξέρετε τους χρόνους για την κατάθεση των τροπολογιών, τροπολογίες μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους κοιόζους εισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Παντσέρη. Είναι πολύ καλή βάση, πολύ καλή έκθεση του κυρίου Παντσέρη για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ όλους. Να κάνω τώρα την ακρόαση για τα βασανιστήρια. Επίσης ένα άλλο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 Vamos a empezar rápidamente nuestra audición sobre... Θα αρχίσουμε την ακρόαση για την 30η επέτειο της ε, Σύμβασης για τα Βασανιστήρια. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να δώσω λοιπόν το λόγο στους ομιλητές μας που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα. Τους ευχαριστώ πολύ που, πήραν, ε, που είναι παρόντες. Ο κύριος Κάστεν Στάουν, που είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος της Δανίας ε, έναντι των Ηνωμένων Εθνών στην ε, Γενέβη. Η Δανία έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση στον αγώνα κατά των βασανιστήριων και μπορεί να μας εξηγήσει πρωτοβουλίες. Και μετά θα έχουμε την κυρία Λάουρα Δολτσικάνα αν προφέρω καλά το όνομά της. Ο κύριος τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να ε, παραστώ εδώ σήμερα και να μιλήσω για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ε, αυτή τη χρονιά. Στις 10 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε την 30η επέτειο της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ της Σύμβασης κατά των βασανιστήριων και είναι σαφές ότι ήταν ο καρπός ε, πολλής και σκληρής δουλειάς ε, από το 1948 όταν ε, θεσμοθετήθηκε ε, η απαγόρευση των βασανιστήριων. Τα πράγματα όμως δεν πηγαίνουν πολύ καλά όχι τόσο καλά όσο θα έπρεπε και βλέπουμε δημοσκοπήσεις που καταδεικνύουν ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά για παράδειγμα τη χρήση βασανιστήριων ε, σε ανακρίσεις ή τέλος πάντων σε προσπάθεια άντλησης πληροφοριών από κάποιον ε, και πολλές φορές αυτά ε, είναι, δημιουργούν παρεξηγήσεις, είναι κάπως παραπλανητικά και στην τηλεόραση και αλλά και σε ορισμένα μυθιστορήματα δράσης. Πολλές φορές ε, λοιπόν τα βασανιστήρια χρησιμοποιούνται όχι μόνο για άντληση πληροφοριών αλλά και για να ε, βλάψει κάποιον, ε, κάποιος κάποιον σωματικά ή συναισθηματικά ή ψυχολογικά να τους υποχρεώσουν να κάνουν πράγματα που κανονικά δεν θα έκαναν και να τους σπάσουν. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε, όπως κάναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ε, την ε, Σύμβαση κατά των βασανιστήριων, ε, την ΟΠΚΑΤ που είναι το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστήριων, τον ειδικό εισηγητή για τα θέματα αυτά, αλλά όλα αυτά είναι πράγματα ρουτίνας. Ε, υπάρχει ένα σύστημα ε, ετήσιο το οποίο όμως ε, δεν καρποφόρησε όσο θα έπρεπε ούτε έλαβε ιδιαίτερη πολιτική όθηση. Ε, γι' αυτό λοιπόν υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία για τη σύμβαση κατά των βασανιστήριων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, χρηματοδότησης ε, του ε, ΟΗΕ για τα θέματα των βασανιστήριων. Θα επανέλθω σε αυτό. Αλλά υπάρχει, και πολιτικά, υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα και ελπίζουμε να μπορέσει η πρωτοβουλία μας να το ανατρέψει αυτό. Ε, υπάρχει πρόβλημα και με την επικύρωση και με την ε, πραγματική εφαρμογή ε, της Σύμβασης κατά των βασανιστήριων. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι είναι μια νέα διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ Δανίας, Μαρόκου και πολλών άλλων χωρών. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι είναι ένα διαπεριφερειακό θέμα. Προσπαθήσαμε να το εξετάσουμε με πολύ επικοδομητικό τρόπο και υπήρξε τεράστια αλλαγή σε σχέση με τα, την συνηθισμένη ε, προσέγγιση που είναι ε, η, καταδίκη, ε, η, η καταδίκαση των βασανιστήριων, το να υπάρξουν επικρίσεις, να υπάρξουν πολιτικές δηλώσεις που επικρίνουν τις χώρες που χρησιμοποιούν βασανιστήρια. Το θέμα όμως είναι ότι όταν βλέπει καλή, κανείς σήμερα τι αποτελεί βασανιστήριο είναι, είναι ένα θέμα αστυνομικής ε, συμπεριφοράς, ε, το θέμα ε, της κράτησης των ανθρώπων που κρατούνται, το πώς γίνεται η μεταχείριση των ανθρώπων και στις φυλακές αλλά και σε ψυχιατρικές κλινικές όταν για παράδειγμα κάποιος έρχεται σε επαφή με μία αρχή και δεν μπορεί να φύγει παρά το ότι απειλείται, πρέπει να ε, δεχθεί την ε, αντιπαράθεση με την αρχή που είναι απέναντί του. Και μερικές φορές ε, υπάρχει κακομεταχείριση, μερικές φορές υπάρχει βασανιστήριο. Πάντως είναι κάτι το οποίο οι δημόσιες αρχές πρέπει πραγματικά να λάβουν υπόψη σε πολλές περιπτώσεις ε, μεταξύ των χωρών ε, που είναι κλειστοφοβικές και που δεν έχουν ε, επικυρώσει ούτε τη σύμβαση ούτε το προαιρετικό πρωτόκολλο δεν είναι θέμα πάντοτε πολιτικής βούλησης. Είναι ένα θέμα σε κάποιο βαθμό του κατά πόσο ας πούμε θεωρεί κάποιος ότι τον ξεπερνούν κάποιες προκλήσεις και ε, το ότι πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια τα οποία δεν μπορεί εύκολα να τα ξεπεράσει. Υπάρχει η αστυνομία και η συμπεριφορά της, η έλλειψη κατάρτισης, η έλλειψη πόρων σε αστυνομικέ δυνάμεις, ε, υπάρχει επίσης το θέμα των εγκαταστάσεων κράτησης. Αν πάει κανείς για παράδειγμα σε διάφορες φυλακές βλέπουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ε, κακές συνθήκες ε, ε, κράτησης. Το όλο θέμα λοιπόν της κράτησης στις ψυχιατρικές κλινικές, για παράδειγμα, ακόμα και στη Δανία, ήταν αντικείμενο δημόσιας κριτικής. Είναι ε, στοιχεία που πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Προσπαθούμε να έχουμε μια θετική προσέγγιση, να λέμε στις χώρες, αν βλέπετε πρόβλημα στην, ε, στο να ξεπεράσετε κάποια εμπόδια, υπάρχουν πράγματα που μπορεί η διεθνής κοινότητα να κάνει για να σας βοηθήσει. Αυτή η προσέγγιση ήταν θεωρούσαμε ότι είναι μια συνεργασία ομοτήμων για να το πω έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν όσον αφορά την βοήθεια προς τις χώρες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά, αλλά σε μερικές περιπτώσεις όταν βλέπουμε για παράδειγμα τις φυλακές ή την αστυνομία, ε, είναι σαν να υπάρχει ένα μαύρο κουτί ε, στις χώρες αυτές. Είναι επιφυλακτικές, δεν θέλουν να, να είναι ανοιχτές σε κριτική, ε, σε μια πιο δυτική προσέγγιση. Είναι πολύ πιο άνετες να μιλούν με γειτονικέ χώρες, ε, ένα μικρό νησί στον Ειρηνικό δεν θεωρεί ότι έχει πολλά κοινά με εμά όσον αφορά ε, τη συνεργασία, για παράδειγμα, με τη Δανία, με μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούν όμως να ε, μάθουν ε, από τι εμπειρίε των υπολείπων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα επικυρώσουν τις την, την σύμβαση αυτή των βασανιστήριων. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους επηρεάσουμε σε σχέση με την απόφασή τους, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα και να εμπνεύσουν και άλλους να προβούν στην επικύρωση. Ε, η στενή συνεργασία λοιπόν μεταξύ γειτόνων είναι σημαντική και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ε, κινητοποιήσουμε πολλούς σε τοπικό επίπεδο στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, ε, στην Ασία αλλά και στην Ευρώπη και επικεντρωνόμαστε στην ευρύτερη ε, Ευρώπη, 54-55 χώρες και χώρες του, χώρες του ΟΑΣΕ ε, ας πούμε, ε, οι οποίες, τους οποίες ζητούμε να προ... υπογράψουν τις δεσμεύσεις αυτής της σύμβασης και του προετικού πρωτοκόλου αυτής. Αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν αποτελεί τη βασική μας προσπάθεια. Ελπίζουμε αυτή τη θετική προσέγγιση να μπορέσουμε να τη δρομολογήσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ διπλωματική δουλειά που πρέπει να γίνει και είναι ένας από τους λόγους που χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Είναι σημαντικό αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορέσει να πιέσει ε, και να ε, προωθήσει αυτή την προσέγγιση ώστε να ε, μπορέσουμε από κοινού να κινητοποιήσουμε πολιτική βούληση αλλά και πόρους προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα... Ε, ε, ε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα Google Friends στη Γενέβη, μια ομάδα φίλων για να αρχίσει να ισχύει το ε, πρόγραμμα εργασίας, το οποίο θα ολοκληρώσουμε κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες, το 2015 θα είναι το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής του προγράμματος. Δεν θέλω να μακρηγορώ, θα ήθελα όμως ακόμη να πω το εξής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε την επίσημη έννοια της επικύρωσης ε, ε, της ΟΠΚΑ, ε, του Προεδρικού Πρωτοκόλου, ως δυνομικό πολιτικό μέσο για την ε, καταπολέμηση των βασανιστήριων. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να πιέσουμε τις χώρες να προσχωρήσουν στη σύμβαση με όσο το δυνατόν λιγότερες επιφυλάξεις, να δεχθούν με μενωμένες καταγγελίες, ε, να κάνουν την παρακολούθηση και να υπάρξει αυτός ο πραγματικός διάλογος με την Επιτροπή κατά των βασανιστήριων και να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις Επιτροπής αυτής. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες ε, μεταγραφής μιας διεθνούς προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο και μπορούμε να το κάνουμε αυτό ενθαρρύνοντας τις χώρες, ε, προσπαθώντας να τους δώσουμε τα μέσα μέσα να το πράξουν και ελπίζουμε ότι έτσι τα αποτελέσματα θα είναι περισσότερο, ε, να είναι πιο σημαντικά από το να ε, καταδικάζουμε απλώς και να χρησιμοποιούμε περισσότερο το μαστίγιο και λιγότερο το καρότο. Το θέμα είναι πώς Κάνουμε τη μέτρηση τώρα των αποτελεσμάτων. Θα, προσπαθούμε να έχουμε, να προσπαθήσουμε να ε, καταρτήσουμε ένα σύστημα δικτών, να υπάρχει τέλος πάντων ένα σημείο αναφοράς μέχρι το τέλος του 2014 ε, κάποιοι δείκτες βάσει των οποίων να μπορούμε να κρίνουμε πόσες ε, ε, χώρες ε, έχουν επικυρώσει, πόσες χώρες έχουν σκοπό να επικυρώσουν και ούτω καθεξής. Έχουμε τουλάχιστον 35 χώρες οι οποίες πρέπει να το κάνουν, αλλά αυτό όμως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η εφαρμογή. Πώς γίνεται η πολιτική επικύρωση να μεταφραστεί σε ε, πράξη σε εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό θέλουμε να παρακολουθούμε να δούμε τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο για να μπορέσουμε να τονίσουμε αρνητικές εξελίξεις σε διάφορες χώρες αλλά και τις θετικές και θα τα αφήσουμε στους υπόλοιπους. Εμείς θα δούμε κυρίως τις θετικές εξελίξεις, τις αρνητικές θα τις δουν οι άλλοι, είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Πιστεύουμε όμως ότι πραγματικά είναι η σωστή προσέγγιση, η θετική προσέγγιση για τα επόμενα δέκα χρόνια δεν ε, αποκλείεται να επιτύχουμε πλήρη επικύρωση από όλες τις χώρες. Η μόνη σύμβαση που μοιάζει είναι η σύμβαση για τα δικαιώματα των ε, παιδιών. Μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Σομαλία δεν έχουν επικυρώσει και ξέρω ότι η Σομαλία πρόκειται να την επικυρώσει αυτή τη σύμβαση. Άρα μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε θα είναι οι χώρες, η χώρα που δεν θα έχει ε, επικυρώσει αυτή τη σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών. Ένα θέμα σαν, το, τα πασανιστήρια που απαγορεύονται από το 48. Ε, είναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ε, πρέπει να ε, εξαλείψουμε αυτό το πρόβλημα. μπορούμε να πετύχουμε πλήρη επικύρωση και θα προσπαθήσουμε για τα επόμενα 10 χρόνια να εργαστούμε πολύ σκληρά γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Στόρ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ντότζι Κάναν της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών υπεύθυνη για τα ανθρωπιστικά ταμεία και το Θελοντικό Ταμείο για τα θύματα της, ε, των βασανιστήριων. Και θα δούμε πριν της δώσω το λόγο ένα σύντομο βίντεο όπου φαίνεται η σημασία της βοήθειας που δίνουν αυτά τα ταμεία. Παρακαλώ.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 to, to the safe place. We feel that our work is, is worth. Our work is never end. Muy bien, muchísimas gracias. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το για αυτό το βίντεο. Είναι μια αγωνίστρια που έχει δώσει πολλά στον αγώνα για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ευημερία των ατόμων, ενώ η ίδια είναι επίσης θύμα, γιατί έχασε τον σύζυγό της σε μια επίθεση κατά της έδρας των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ. Οπότε θέλουμε να αποτίσουμε και ένα φόρο τιμή ε, και στα θύματα όλων αυτών των επιθέσεων. Ευχαριστούμε πολύ για την εργασία σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Είναι τιμή και χαρά η παρουσία μου εδώ εξ ονόματος ε, του είπα προσώπου Ανθρωπέων δικαιωμάτων στη Γενέβη. Νομίζω ότι οι εικόνες και τα λόγια ήδη μίλησαν από μόνα τους. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε ο πρέσβης. Την επόμενη εβδομάδα κλείνουν 30 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης κατά των βασανιστήριων. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να καταπολεμήσουν τα ενωμένα Έθνη τα βασανιστήρια. Υπάρχει ένα προεδρικό πρωτόκολλο, υπάρχουν ε, οι θεματοφύλακες αυτής της σύμβασης. Ε, υπάρχει ένας ειδικό συζητητή και υπάρχει και ένα ταμείο για τα θύματα βασανιστήριων. Το ταμείο αυτό υπάρχει εδώ και 33 χρόνια. Το ταμείο υπήρχε, υπάρχει, γιατί υπάρχουν χιλιάδες θύματα βασανιστήριων που βρίσκονται στο περιθώριο σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Και πραγματικά χαιρετίζω την έμφαση που δόθηκε στην επικύρωση και στην εφαρμογή, γιατί αυτό είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τη σύμβαση και το άρθρο 14 που αναφέρει σαφώς ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχει αποκατάσταση των θυμάτων ε, βασανιστήριων. Αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστήριων δεν είναι μία φιλανθρωπική πράξη, είναι μία νομική υποχρέωση που έχει σχέση με ένα εκτελεστό δικαίωμα. Ο αριθμός και μόνον των θυμάτων που προσεγγίζουν το ταμείο μας, καθώς και άλλα ταμεία, είναι εντυπωσιακό. Υπάρχουν και μαρτυρίες που συλλέγονται από την Επιτροπή και λένε από μόνα τους ότι δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτή η υποχρέωση. Το ταμείο έχει μία μοναδική δυναμική. Το ταμείο είναι επικεντρωμένο στα θέματα των, σε θέματα που αφορούν τα θύματα βασανιστήριων. Είναι ένα καινούριο ταμείο, τα Ηνωμένα Έθνη πέρα από τη, με την εξαίρεση το Διεθνές Γραφείο Εγκλημάτων υπάρχει ένα ταμείο για τα θύματα. Εδώ έχουμε ένα ταμείο που παρέχει άμεση βοήθεια στα θύματα. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει στο μηχανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Να δούμε πρακτικά πώς λειτουργεί αυτό το ταμείο. Με την εθελοντική συμβολή δωρητών και των κρατών και διοχετεύει τα χρήματα αυτά σε πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που απευθύνονται απευθείας στα θύματα παρέχοντάς τους ε, ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική, ανθρωπιστική βοήθεια. Σε αυτή την εξίσωση Υπάρχει και η συμβολή των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων γιατί υπάρχει μια ομάδα η οποία συμβουλεύει το Γενικό Γραμματέα σχετικά με την αποκατάσταση και τη χρήση των κονδύλιων και βεβαίως ε, ο υπερός εκπρόσωπος. Με το πέρασμα του χρόνου δόθηκε βοήθεια δίνεται βοήθεια σε 30.000 θύματα το χρόνο σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο επαγγελματιών συμπεριλαμβάνοντας ψυχολόγους, ε, δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν αναπτύξει μία τεχνογνωσία για το πώς παρέχεται βοήθεια στα θύματα των ε, βασανιστήριων. Το Ταμείο βασίζεται, στηρίζεται στην παροχή βοήθεια σε θύματα και θεωρεί ότι είναι μία μακροπρόθεσμη δέσμευση. Τα, οι των βασανιστήριων μπορούν να περάσουν και από τη μία γενιά στην άλλη. Παράλληλα όμως το Ταμείο παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης, όπως σας είπα, τα τελευταία δύο χρόνια ξεκινήσαμε προγράμμα, να εφαρμόζουμε προγράμματα στα σύνορα με τη Συρία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία. Παρέχουμε βοήθεια στους ε, πρόσφυγες με τη βοήθεια του κυρίου Αχμέντα αντιμετωπίζουμε την κρίση στο βόρειο Ιράκ και τους τελευταίους μήνες ξεκίνησε ένα project στην ε, Ουκρανία. Το Ταμείο προσπαθεί να έχει την απαιτή τις απαιτούμενες δυνατότητες για να αντιμετωπίσει τα θύματα, τα καινούργια θύματα. Όπως ε, σας είπα, συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών που παίζει καθοριστικό ρόλο και συμπληρώνει πολύ συχνά τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οργανώσεις ε, κρατικές. Όπως σας είπα υπάρχει το άρθρο 14 της Σύμβασης που καθιστά υποχρεωτικό για το κράτος να παρέμβει. Όταν όμως είναι λιματικό το κράτος παρέχεται, αυτή είναι η μοναδική ε, βοήθεια που παρέχεται στα θύματα και νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε την δέσμευσή τους ε, γιατί πάρα πολύ συχνά αυτό γίνεται εις βάρος ε, με, κίνδυνο της προσωπικής τους ε, ζωής, ε, της ζωής τους. Να σας παραθέσω ένα-δύο αριθμητικά στοιχεία. Δυστυχώς τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρήθηκε μία πτωτική στάση στις δωρεές. Τα τελευταία 30 χρόνια το ταμείο έφτασε σε 150.000 δολάρια, τα οποία τα διοχέτευσε σε διάφορες πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο. Και βοήθησε πάνω από 600 οργανώσεις, ε, ομάδες γιατρών, ψυχιατρικά τμήματα, εξειδικευμένα κέντρα, ομάδες δικηγόρων. Η μορφή της βοήθειας μπορεί να προσλάβει διάφορες ε, το ίδιο βοήθεια βοήθεια μπορεί να προσλάβει διάφορες μορφές. Προσπαθούν να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και το ποσό που θα μας χρειαζόταν, το ιδανικό ποσό, είναι γύρω στα 12 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Φέτος ήμασταν στα 8 εκατομμύρια. Του χρόνου θα στηρίξουμε 109 πρωτοβουλίες σε όλες τις περιοχές του κόσμου και θα διοχετεύσουμε 7 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια. Να σας δώσω μερικά στοιχεία που ενδεχομένως παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. Το Ταμείο το 2015 επενδύσουμε πάνω από ένα εκατομμύριο, 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε 40 έργα που παρέχουν βοήθεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 16 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή των ευρωπαϊκών χωρών ήταν ιδιαίτερα σημαντική για το Ταμείο. Δυστυχώ, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μια πτωτική τάση. Τα προηγούμενα χρόνια 18 χώρες συνέβαλαν. Σήμερα συνέβαλαν μόνο 5 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπρόσωπο της μία εξ αυτών βρίσκεται δεξιά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δανία, η Γερμανία επίσης υποστηρίζει πολύ τις δράσεις μας, η Ιρλανδία, η Φιλανδία και η Αυστρία. Χάσαμε όμως πολλές χώρες καθοδόν. Βεβαίως η οικονομική κρίση έπληξε όλους μας. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη στήριξή σας, η οποία δεν σημαίνει ότι κατά ε, ότι κατά ανάγκη πρέπει να είναι οικονομική, α είναι και πολιτική. Τα βασανιστήρια είναι μία πρακτική που δυστυχώ εφαρμόζεται παντού. Παρόλα ε, όσα ε, συνέβησαν, πάντοτε υπάρχει κίνδυνος συνέχισης των βασανιστήριων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει έντονη παρουσία της τρομοκρατίας ή της αντιτρομοκρατίας που θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν τα βασανιστήρια. Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτή την ευκαιρία για να κάνω ταπεινά μια, ένα αίτημα. Good rehabilitation is an investment for future generations. Είναι λοιπόν καλή επένδυση η καταπολέμηση των βασανιστήριων να αποτρέπει τα βασανιστήρια και διάφορες χώρες έχουν εγκρίνει νόμους για την καταπολέμησή τους. Ένα θύμα που αποκαθίσταται, αποκαθίσταται είναι ήδη κάτι το θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόγμπιλερ. θα αναφερθεί στα βασικά σημεία της έκθεσης πρωτοβουλίας που κάναμε το Μάρτιο στο Κοινοβούλιο και μερικά σημεία για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Πέρυσι η Βερονίκ Ντεκάιζερ είχε συντάξει μια έκθεση που εγκρίναμε λοιπόν, δηλαδή φέτος μέλλον καλύτερα, μάλλον καλύτερα, για την κατάργηση των βασανιστήριων στον κόσμο. Βεβαίω ε, στα λόγια όλοι καταδικάζουν, όλες οι χώρες καταδικάζουν τα βασανιστήρια, αλλά πολύ λιγότερη είναι η πολιτική βούληση για να αναλυφθούν πρωτοβουλίες για την κατάργηση των βασανιστήριων, γιατί σε πολλές χώρες διαπιστώνουμε ότι αυτά τα εγκλήματα και παραβίαση των δικαιωμάτων συνεχίζονται. Το ψήφισμά μας επικρίνει το ότι τα κράτη-μέλη και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν κάνουν αρκετά για να υλοποιήσουν τη δέσμευσή του κατά των βασανιστήριων. βεβαίω έχουμε θαυμάσιες κατευθυντήριε ως Ένωση. Αλλά είναι κενό γράμμα κυρίω. Το Μάρτιο λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες για να εφαρμοστούν αυτές οι οδηγίες και να εμπλακεί περισσότερο το Κοινοβούλιο στην επιτήρηση της πολιτικής. Ίσως θα μας πει περισσότερα η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επίσης καλέσαμε την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να είναι πιο φιλόδοξη για να ε, ε, βοηθάει τους τοπικούς και περιφερειακούς μηχανισμούς αντιμετώπισης και καταπολέμησης των βασανιστήριων. Και ίσως θα μπορούσε να υπάρχει και ένα παγκόσμιο δίκτυο. Δεν έχουμε κάνει πολλά γι' αυτό. Και το ψήφισμα επίσης καλούσε όλες τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και τις πρεσβείες των κρατών μελών να αξιοποιήσουν την Διεθνή Μέρα για τα θύματα των βασανιστήριων 26 Ιουνίου για να προωθήσουν ε, τη βοήθεια προς τα θύματα και να εμπλέξουν και την κοινωνία των πολιτών σε αυτές τις προσπάθειες. Περαιτέρω το ψήφισμα έλεγε πολύ συγκεκριμένα ότι τα κράτη-μέλη, του Κοινοβούλιο και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να κάνουν περισσότερες επισκέψεις σε τόπους κράτησης. Το είπε και ο κύριος Στάρ. Είναι τα αστυνομικά τμήματα, είναι οι φυλακές, τα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Πρέπει να κάνουμε τέτοιες επισκέψεις. Και ξεκινήσαμε και την εκπόνηση ενός ε, πρακτικού οδηγού για τους ευρωβουλευτές για το πώς να επισκέπτονται τόπους κράτησης κατά τις επισκέψεις τους σε διάφορες χώρες. Και να δούμε τι έχει γίνει γι' αυτό. Ακόμη και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισκεφθεί το Αζερμπαϊτζάν να δει ποια είναι η κατάσταση για τη Λάιλα Γιούνους. Πολύ συχνά μας λένε δεν «Ναι, μας επιτράπει να επισκεφθούμε αυτή τη φυλακή. Αλλά πρέπει να έχουμε καταφυντήριες γραμμές ακόμη και για λιγότερο γνωστές περιπτώσεις να έχουμε δυνατότητα να επισκεπτόμεθα τις φυλακές αυτές. Όπου κρατούνται δηλαδή. Και όπως μας είπε και η κυρία Ντόλτζη Κανάντσες, ζητήσαμε να υπάρχουν περισσότερες πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε τα θύματα και να συμβάλλουμε και στη χρηματοδότηση του Ειδικού Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών. Το ψήφισμά μας επίσης ασχολήθηκε ιδίω με τα βασανιστήρια κατά των παιδιών και τη βία με βάση το φύλλο. Όπου νομίζω ότι εκφράσαμε και μια καινούρια αντίληψη ότι η θανατική ποινή είναι αντίθετη με τη Διεθνή Σύμβαση κατά των Βασανιστήριο. Και καλέσαμε την Ένωση να προσαρμόσει λοιπόν την πολιτική της για τη θανατική ποινή. Αυτά λοιπόν είπαμε στην έκθεση, αλλά δεν τα συζητήσαμε κατόπιν στο Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να μας πει λοιπόν η υπηρεσία εξωτερική δράση πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. και να θέσω και μερικές ερωτήσεις. Εφτά λεπτά έχουμε. Νομίζω λοιπόν τότε να ακούσουμε και την άποψη της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για να δούμε τι έχουν κάνει για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να δώσω πρώτα τον λόγο στους δύο προσκεκλημένους μας, αν θέλουν να απαντήσουν. Και αν έχουμε χρόνο θα δώσουμε και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ο κύριος Τόου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ διάβασα προσεκτικά τη δήλωση του Κοινοβουλίου του Μαρτίου του τρέχοντος έτους και μου έκανε πολύ εντύπωση η διεξοδική ανάλυση και η διατύπωση της συγκεκριμένης δήλωσης. Μερικά, μερικές σκέψεις μου για να είμαστε αξιόπιστοι για το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάποια γνώση ότι το βασανιστήριο δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι που συμβαίνει και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ μερικές φορές. Στα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, ε, πριν από μερικά ε, χρόνια είχαν, είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας κάποια πολύ κακή μεταχείριση ετούντων άσυλο σε μερικά κράτη-μέλη. Είναι αυτά λοιπόν ζητήματα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερο ρόλο να διαγραμματίσει στο, στις χώρες που είναι εντό, κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κάφκασο, ε, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα διαλόγου με αυτές τις χώρες και ως μέλος αυτής της διαπεριφερειακής ομάδας ε, χωρών έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βέβαια και άλλοι να ε, κινητοποιήσουμε ε, κάποιες προσπάθειες στις χώρες αυτές. Όπως επίσης ε, και στη Λατινική Αμερική, στη Μέση Ανατολή υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνουμε καλά ως Ευρωπαίοι και πράγματα που κάνουμε λιγότερο καλά. Μερικές φορές θεωρούμαστε εισβολέας και όχι ευπρόσδεκτος προσκεκλημένος. Και αυτό το είπα και στην εναρκτήρια ομιλία μου. Πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα σε γειτονικέ χώρε που έχουν αντιμετωπίσει ε, τέτοια προβλήματα και που θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα, αλλά από γειτονικέ χώρε και όχι τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό. Είναι δύσκολο το όλο θέμα τη μεταχείρισης των φυλακισμένων, των ε, ε, ανθρώπων που είναι σε ψυχιατρικέ κλινικέ, των ανθρώπων που έχουν έρθει σε επαφή με αστυνομία. Μιλάμε για ανθρώπους ε, που είναι το βασικό μας μέλημα. Οι πολιτικές ευαισθησίες είναι σημαντικές στη διπλωματία και πρέπει να δουλεύουμε με χώρες, ε, να συνεργαζόμαστε με χώρες που πρωτοστατούν στην περιφέρειά τους. Είναι καλύτερο να κάνουμε αυτό από το να είμαστε ένας εντελώς ξένος παράγοντας που φαίνεται σαν να προσπαθεί να ε, εισχωρήσει στα δικά τους. Ε, υπάρχει και πολιτικός ρόλος τον οποίο μπορούμε να διαδραματίσουμε, μπορούμε να πιέσουμε, μπορούμε να τονίσουμε, μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις πολιτικής, μπορούμε να υποστηρίξουμε τοπικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα θέματα αυτά. Ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και πότε να ε, κάνουμε στην άκρη και να τα αφήσουμε σε άλλους ε, να βοηθήσουν μια χώρα να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ντόλτσι Κανάν. Ευχαριστώ πολύ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπε μόλις ο κύριος Στάουρ είναι πάρα πολύ περιεκτική η δήλωσή σας πράγματι και κατά την άποψή μας ε, ε, πολύ καλά κάνετε και τονίζετε ιδιαίτερα διάφορες ε, ομάδες στόχο, ομάδες που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν όλο και περισσότερες γυναίκες θύματα ε, και το ακούμε, το βλέπουμε από τις διάφορες αιτήσει. 56.000 ε, είναι ε, τα θύματα, 26.000 θα είναι γυναίκες βάσει των στατιστικών μας. Νομίζω λοιπόν ότι τα... Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και συνεπώς η, η η έμφαση που δίνεται ε, στους, ε, στα ομοφιλοφίλους, στις γυναίκες και στα παιδιά είναι πάρα πολύ σωστή. Ε, επίσης πάρα πολύ, καλά ζητάτε, πάρα πολύ σωστά ζητάτε χρηματοδότηση, η αποκατάσταση αλλά και η πρόληψη είναι σημαντική. Μη, είπατε ότι υπάρχει, είπαμε ότι υπάρχει ένα ειδικό ταμείο ε, του προαιρετικού πρωτοκόλου 230.000 ε, δολάρια σε εισφορές έλαβε σήμερα και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στην αρχιτεκτονική της πρόληψης. Καλύτερα να μην το σκοτώσουμε ε, πριν γεννηθεί καν. Ελπίζουμε λοιπόν ότι στο επόμενο σχέδιο δράσης ε, θα διατηρηθεί η έμφαση στα βασανιστήρια και να είναι τόσο ισχυρή έμφαση αυτή όσο και η διατύπωση που χρησιμοποιήσατε στο ψήφισμά σας. Bueno, por dos minutos y creo que ya sin interpretación porque ha concluido el tiempo de los. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμη λεπτά και μετά οι διερμηνείς θα πρέπει να αποχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, mais on m'avait écrit votre prénom en anglais, alors j'ai imaginé que votre nom était aussi en anglais.